Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο σημαντικότερος συνάδελφος για την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόν. Είναι ο συνάδελφος εισηγητής, έτσι λοιπόν μπορούμε να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Βεβαίω μας έδωσαν μια καταπληκτική αίθουσα, πολύ βολική, στο κέντρο του Κοινοβουλίου, αλλά δυστυχώς αν παραμείνει τόσο άδεια όσο είναι τώρα, πρέπει να σας πω τελείως ειλικρινά ότι δεν θα μπορέσουμε να την κρατήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ας πάμε, εν πάση περιπτώσει, στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Το πρώτο θέμα, όλα είναι πολύ σημαντικά τα θέματα, αλλά εδώ πρόκειται για μια δική μας ε, έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής ε, Ήτρε. Η συγκεκριτής είναι ο από το ΕΛΚ, από τη Λιθουανία και Έχετε καταθέσει 821 τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης του κυρίου Σαουντάργας και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι σκιώδεις εισηγητές, εξ όσων γνωρίζω, θα συναντηθούν αργότερα σήμερα για να συμφωνήσουν τουλάχιστον στις ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες. Έχουμε μία ώρα για τη συζήτησή μας, ίσως και λιγότερο, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να ψηφίζουμε ακριβώς στις 10 η ώρα. Και ελπίζω τότε να έχουν έρθει όλα τα μέλη και τουλάχιστον η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Αν ε, λοιπόν ε, κάποιος ε, θέλει να δει πώς είναι στην αίθουσα να το ρίξει στι 10 η ώρα. Συνάδελφε Σαντάρκας, έχετε το λόγο και παρακαλώ να μιλήσετε για 5 περίπου λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που δώσατε τόσο μεγάλη σημασία στην έκθεσή μου. Με 821 τροπολογίες αυτό καταδεικνύει ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει εδώ και πολύ καιρό στη δική μας την ημερήσια διάταξη, στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται σχεδόν κάθε μέρα. Είναι κατανοητή λοιπόν ε, η σημασία που το αποδίδεται. Και επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες ε, γενικές, ε, γενικής φύσεως παρατηρήσεις όσον αφορά τη στρατηγική μας για τις τροπολογίες. Βεβαίως και προσπαθούμε να ε, λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις ε, παρεμβάσεις αλλά δεν είναι δυνατόν να δώσουμε την ίδια σημασία σε όλες τις τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα βασικά θέματα. Και κάποιες ε, δευτερευού σημασία τροπολογίες αναγκαστικά θα παραμεληθούν περισσότερο σε σύγκριση με τις άλλες. στο Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, το βασικό καθήκον μας είναι να επεξεργαζόμαστε, να επιδιώκουμε την βαθιά και ευρεία συνένεση των πολιτικών κομμάτων για τα θέματα που συζητάμε. Ε, και γι' αυτό συζητούνται ε, πολλές φορές τα θέματα που μας απασχολούν. Και κάτι άλλο, μια επίσης γενικής φύσης παρατήρηση που μπαίνει όμως στην ουσία του θέματος στην αρχή μιλάμε για την Ενεργειακή Ένωση. Η Ενεργειακή Ένωση, Ένωση ε, θα παρουσιαστεί και αύριο. Μιλάμε λοιπόν για ένα μετακινούμενο στόχο που είναι η Ενεργειακή Ένωση, που όμως ο στόχος αυτός έχει ήδη φτάσει. Άρα δηλαδή θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτήν την έκθεση. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι όσον αφορά στις τροπολογίες πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ε, ενεργειακή ασφάλεια στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης. Και βεβαίως και υπάρχουν άλλα θέματα που μπορεί κανείς να συζητήσει σε σχέση με την Ενεργειακή Ένωση. Αυτό ήθελα να το προτάξω ως πρώτη μου παρατήρηση. Τώρα, μία δεύτερη παρατήρηση που αφορά, αφορά στην ενεργειακή επάρκεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι όλοι σας γνωρίζετε ότι η ενεργειακή επάρκεια είναι πολύ σημαντική ε, θα εξετάσουμε λοιπόν τις ε, τροπολογίες ε, κάτω από το πρίσμα της ενεργειακής επάρκειας και θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε όσο δυνατόν περισσότερες τροπολογίες που αφορούν στην ενεργειακή επάρκεια. Παρόλα αυτά όμως η ενεργειακή επάρκεια δεν είναι ο απόλυτος στόχος. Υπάρχει μία ρίση ότι η καλύτερη ενέργεια, η καλύτερη μορφή ενέργειας είναι αυτή που δεν χρησιμοποιείται. Αυτό είναι εντυπωσιακό άποψη, αλλά ξέρετε, αν δεν υπάρχει πρόσβαση στην ενέργεια, τότε τι είδου επάρκεια θα υπάρχει. Βεβαίως και η ενεργειακή ασφάλεια συμβαδίζει με την ενεργειακή επάρκεια. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε στην εκθεσή μας όσο δυνατόν περισσότερο την ενεργειακή επάρκεια. Όσον αφορά τώρα την εγχώρια ενεργειακή παραγωγή, υπάρχει το ενεργειακό μείγμα. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως, από την άλλη, τα κράτη-μέλη οφείλουν να επεξεργάζονται την προσέγγιση τους ε, μέσα από το συντονισμό και μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και εδώ πρέπει να αναζητήσουμε το συμβιβασμό. Ε, που δεν ή δεν μπορούμε να υπογραμμίζουμε ή να θέλουμε να προβάλλουμε ότι στόχος είναι μπορουμε να υπογραμμιζουμε η να θελουμε να προβαλλουμε οτι στοχος ειναι η μειωση ο περιορισμό αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι να καταλήξουμε σε μία προσέγγιση και τέλος αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εξωτερική διάσταση του θέματος. Στη δική μας την έκθεση αναφέρουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω στις ε, μεθόδους προσέγγισης και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί μια συγκεκριμένη στρατηγική πώς είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να ε, βλάψει την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών ή οτιδήποτε παρεμφερές. Άρα δηλαδή ήδη υπάρχουν πολλά θέματα που χρήζουν συζήτηση. Προσβλέπω με χαρά στη συζήτηση με τους εσκιώδεις εισηγητές αλλά και με όλους τους άλλους συναδέλφους για να επιδιώξουμε ένα ως το δυνατόν βαθύτερο και ουσιαστικότερο συμβιβασμό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και εμείς συνάδελφε ο συνάδελφος Πόχε ε, έχει το λόγο σε σκιώδης εισηγητής εκ μέρους των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή για το έργο του. Ε, πρέπει να ήταν πολύ περίπλοκη δουλειά με πάνω από 800 τροπολογίες. Αυτό βέβαια καταδεικνύει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και αυτός ο μεγάλος αριθμός ε, τροπολογιών απλώς το επισημαίνει περαιτέρω. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι κάτι περίπλοκο και χαίρομαι που η συζήτησή μας δεν περιορίζεται μόνο ε, στα ορυκτά καύσιμα όπως ε, είχε φανεί αρχικώς, αλλά εξετάζουμε γενικότερα το ζήτημα. Οι συμβαστικές προτάσεις αποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε μόνο υπόψη ε, τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, αλλά θα πρέπει αυτές να ενταχθούν και σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Οι τροπολογίες που υπευλήθησαν ε, αποδεικνύουν ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι καταρχάς ε, δική μας ευθύνη και προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια, θα πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όχι μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και σε επίπεδο εθνικής πολιτικής των κρατών μελών. Είμαι ε, πάρα πολύ ευχαριστημένος, διότι στις συμβιβαστικές προτάσεις αναφέρονται θέματα όπως η ενεργειακή απόδοση, ε, διότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια. Θεωρώ ότι στη διάρκεια του απογεύματος, ε, στη συνεδρίαση με τους κοιόδης εισηγητές, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αρκετούς συμβιβασμούς, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε και μια λύση για όλες αυτές τις τροπολογίες. Υπάρχουν κάποια θέματα ε, τα οποία θα ήθελα να θίξω, ε, ιδίως όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και την ενεργειακή απόδοση. Είναι θέματα στα οποία θα ήθελα να σταθούμε λίγο παραπάνω, αλλά έχουμε σίγουρα θετική στάση. Ευχαριστώ πολύ, ε, συνάδελφε. Ο Άσλι Φόξ, εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχά, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τι συμβιβαστικέ προτάσει. Με τόσο πολλέ τροπολογίε που επευλήθησαν, ε, αντιλαμβάνομαι ότι θα του πήρε πάρα πολύ χρόνο. Δυστυχώ, το γεγονός ότι έχουμε τόσε πολλές τροπολογίες που ζητούν τόσο πολλά μεμονωμένα μέτρα μα ε, μας οδηγεί ίσως ε, στον κίνδυνο να χάσουμε την ουσία αυτή τη έκθεση. Δεν θέλουμε ένα χριστουγεννιάτικο ε, δέντρο στο οποίο καθένα θα έχει κρεμάσει τη δική του χρωματιστή μπάλα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή στάση ως προς το τι μπορούμε να επιτύχουμε και πώς μπορούμε να έχουμε μια λογική έκθεση από τον εισηγητή, διότι αυτό θα συνεισφέρει ε, τα μάλλα στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του ζητήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, φαίνεται, να αυξήσουμε τη διασύνδεση και να ολοκληρώσουμε την ε, ενεργειακή αγορά. Αυτό θα μας οδηγήσει τελικά σε ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, πολύ σωστά ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους αρμόδιους φορείς να δράσουν υποστηρίζοντας έργα υποδομών, για παράδειγμα, κοινού ενδιαφέροντος αλλά όπου είναι δυνατόν θα πρέπει να επιμείνουμε στις ευρύτερες αρχές και να αποφύγουμε τις περιττές λεπτομέρειες. Θα πρέπει να επισημάνουμε πού θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα ώστε να έχουμε νέα αγορά, ώστε σύν χρόνο να μπορέσουμε να ε, αφήσουμε την ενεργειακή νέα αγορά να λειτουργήσει. Σε 10 χρόνια θα πρέπει να είμαστε σε θέση ε, αν ο Πούτιν αποφασίσει να κλείσει όλε τι τρόφιγγε φυσικού αερίου, να μην μα νοιάζει, γιατί η Ενεργειακή μα Ένωση θα μα παρέχει φυσικό αέριο από άλλε πλευρέ. Καλωσορίζω βέβαια και τις διάφορες εκκλήσεις ε, στη συμβαστική πρόταση να διασφαλίσουμε πλήρη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας από όλα τα κράτη-μέλη, κυρίως στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια. Και επίσης καλωσορίζω και την, ο γεγονός ότι ε, καλούμαστε να ληφθεί υπόψη η τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, ώστε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τις, ε, τους ίδιους πόρους ενέργειας όταν θα αναπτύσσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια. Θα πρέπει βέβαια να προσέξουμε κάποια στοιχεία. Η συμβαστική πρόταση παράγραφη 6 για παράδειγμα, όπου λέγεται ότι η ε, απομάκρυση του άνθρακα από το ενεργειακό μείγμα είναι πολύ σημαντικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε στη σημασία της ε, τεχνολογικής ουδετερότητας και τη σημασία της αγοράς στη μία παράγραφο και μετά στην επόμενη παράγραφο να λέμε ότι το ενεργειακό σύστημα θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν θα βασίζεται και σίγουρα όχι για τις περισσότερες χώρες και επίση δεν εξαρτάται από εμά. Το ενεργειακό μείγμα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επίσης, αναφερόμαστε στην ανάγκη έγκριση και έγκαιρης εφαρμογής της οδηγίας NIS και του ε, πακέτου ε, των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεν ξέρω από πού θα προέρθουν. Αυτά είναι θετικά στοιχεία μεν, αλλά δεν αποτελούν την πλήρη απάντηση και δεν θα πρέπει να κρυφτούμε πίσω από αυτά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα για την ασφάλεια και η χρηματοδότηση θα πρέπει να προκύψει και από άλλε πηγέ και όχι από την ανακατανομή του ευρωπαϊκού προπολογισμού από πολύ σημαντικέ μάλιστα πηγέ όπω για παράδειγμα η έρευνα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος και ο δυσυγητής εξ στο των φυσιλελευθέρων, ο κύριος Πέτερσεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή, καταρχάς, για την πολύ μεγάλη δουλειά που έκανε να πω ότι δεν το ζηλεύω καθόλου τον εισηγητή που χρειάστηκε να συνδυάσει όλες αυτές τις τροπολογίες, αλλά χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει τόσο πολύ υλικό ε, και υπάρχουν πολλά στοιχεία κοινά και χαίρομαι τουλάχιστον διότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια κοινά σημεία σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια βασικά στοιχεία και τροπολογίες ε, που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ε, κυβερνοασφάλεια έχουμε υποβάλει μια τροπολογία, την 166, η οποία επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι τα ΕΦΗ e δίκτυα και τα ενεργειακά δίκτυα θα προστατεύονται από ε, τι ολοένα και πιο υψηλής τεχνολογίας επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που έρχονται από όλε τι μεριέ του κόσμου. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ε, δώσουμε μια εύρωστη απάντηση για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε κάποια κοινά σημεία, να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα μέσα για να αντιμετωπίσει αυτέ τι προκλούσει. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα, αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλη χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτέ τι πολύ επικίνδυνε προκλήσει. Δεύτερον, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, που είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα για όλου μα. Ε, θα ξεκινήσουν οι προτάσεις για την Ενεργειακή Άνωση ε, αύριο επισήμως και ε, είναι σαφές ότι η ενεργειακή ασφάλεια εξαρτάται από όλους εμάς και από τη συνεργασία μας, η οποία θα πρέπει να αυξηθεί και ε, επιπλέον θα πρέπει να τηρήσουμε και τις υποχρεώσεις μας, να εφαρμόσουμε πλήρως τις, ε, την κείμενη νομοθεσία, κυρίως την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια. Επίσης, πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, και ε, θέλουμε να τονίσουμε και πόσο σημαντικό είναι να συμμορφωθούμε με τους στόχους της ενεργειακής απόδοσης ε, για το θέμα αυτό και να μειώσουμε τη συνολική μας κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες που έχουν επιβληθεί προς αυτό το σκοπό και ελπίζω να μπορέσουμε να τις εξελίξουμε περαιτέρω, κυρίως την 315. Ε, Από την οικονομική σκοπιά τώρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το σχέδιο Juncker θα έχει αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχουν πάρα πολλά ιδιωτικά κονδύλια και ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλά έργα. Ε, εξελίξει. Η πρόκληση είναι πώς να ενώσουμε όλες αυτές τις τελίτσες. Πώς να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και να ε, έχουμε έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μορφή χρηματοδότησης που θα διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο και τις υποβολές αιτήσεων, αλλά και την έγκριση αυτών των ε, προγραμμάτων για επιχορήγηση. Ένα σταθερό λοιπόν ρυθμιστικό πλαίσιο γι' αυτό θα μας διασφαλίσει ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλή ε, χρήση των κεφαλαίων και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Και να σας επισημάνω και την τροπολογία 206, την οποία θα θέλαμε να ε, έχουμε και να εξελίξουμε περαιτέρω. Τέλος, η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι πολύ σημαντική και ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες που υπευλήθησαν προς αυτό το σκοπό. Θα θέλαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να τονίσουμε πόσο πολλές ευκαιρίες υπάρχουν θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς ε, σε όλον αυτόν τον κλάδο, για παράδειγμα ενεργειακή απόδοση, ευφυείς τεχνολογίες. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ <clears throat> για τις παρατηρήσεις σας ε, εκ μέρους της Άλτη και τώρα εκ μέρους των Πρασίνων, κύριο Γιάβο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το τιτάνιο έργο του και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. φαίνεται ότι έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε σχεδόν πλήρως σε πολλά ζητήματα, για παράδειγμα την ενεργειακή αποτελεσματικότητα ε, και άλλα θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Σε αυτά τα θέματα υπάρχει συμφωνία. Και αυτό νομίζω υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Τα εξής. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις και κάποια επιμέρους ζητήματα που οι πράσινοι τα θεωρούν σημαντικά. Όταν υποβάλαμε τις τροπολογίες μας, είπαμε ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα ε, ευχολόγιο, δεν πρέπει να έχουμε συστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να μετρηθούν. Αντιθέτως, χρειαζόμαστε συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένα μέτρα. Δεν βοηθά να συνεχίσουμε να καταγράφουμε σε ένα χαρτί ε, τις επιθυμίες μας χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα τις επιτύχουμε, πώς θα τα επιτύχουμε όλα αυτά. Και με αυτή τη λογική συντάξαμε τις τροπολογίες μας προσπαθώντας να ε, υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας και παλαιότερες θέσεις που έχει ε, υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με διάφορα έγγραφα, με διάφορα ψηφίσματα σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια καθώς επίσης και τους στόχους για την ε, κλιματική αλλαγή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την, αποτελεσμα... αποτελεσματικότητα και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ε, επιμείνουμε σε αυτέ τι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην επιτρέψουμε ούτε στο Συμβούλιο ούτε στην Επιτροπή να υπονομεύσει τι θέσει που έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο επανειλημμένα. Γι' αυτό λοιπόν παραπέμπουμε σε προηγούμενα ψηφίσματα και προηγούμενε αποφάσει του ε, Κοινοβουλίου στην στρατηγική. Δεύτερη γενική παρατήρηση. Είναι σημαντικό η στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια να ταιριάζει με τις υπόλοιπες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι ε, μεμονωμένο, ξεχωριστό πρέπει να είναι συνεχτική με τις υπόλοιπες πολιτικές και στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για παράδειγμα την ε, στρατηγική και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Είναι ουσιώδους σημασίας να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της ενεργειακής στρατηγικής και τους στόχους που έχει αποδεχθεί και έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Και τώρα περνώ στα επιμέρου. σας υπόσχομαι κύριε Πρόεδρε δεν θα με ακρηγορήσω. Οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι πολύ σημαντικό θέμα και χρειάζονται μέτρα για αυτέ για να έχουμε στην Ευρώπη ε, αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική. Τώρα υπάρχει το ζήτημα της ενοποίησης των αγορών, όχι μόνο στο επίπεδο των υποδομών, αλλά επίσης και στο νομικό, στο ρυθμιστικό, καθώς επίσης και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, τα εφή δίκτυα, Χρειάζεται λοιπόν ε, διασύνδεση και στο τεχνολογικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των ρυθμιστικών αρχών. Επίσης είναι σημαντική, σημαντικό να είναι ε, ε, φτηνή η ενέργεια και να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από εξωτερικούς παρόχους, όχι μόνο από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, αλλά και γενικότερα. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα εκ μέρους της ΓΚΟΕ ακριβώς δίπλα ε, ο κύριο Νεοκλής Σιλικιώτης, ο οποίος είναι και σχεδόν εισηγητής. Παρακαλώ. Στον Πρόεδρε. Ε, πρώτα να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Σαουδάρκας. Ε, έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά και θεωρώ ότι είναι σημαντικό το βήμα που γίνονται με τις συμβαστικές προτάσεις. Όμως στην έκθεση υπάρχουν ορισμένα κενά που πρέπει να συμπληρωθούν. Αρχικά είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η ανάγκη ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια απορρέει από το γεγονό ότι η ενέργεια συνιστά βασικό ανθρώπινο αγαθό στο οποίο πρέπει όλοι έχουν πρόσβαση. Προ αυτήν την κατεύθυνση χαιρετίζομαι την αναφορά που προτείνεται στι συμβαστικέ τροπολογίε όσον αφορά την ανάγκη να καταπολεμηθεί το νέο φαινόμενο τη ενεργειακή στόχια. Εν τούτης είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εν λόγω παράγραφος. Το δεύτερο πρέπει να τοριστεί περαιτέρω η ανάγκη άμεση πρόθεση μέτρων για άρση τη απομόνωση κρατών ή και περιεχών από τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα. Είναι γνωστό ότι υπήρχε ένα στόχο που έχει τεθεί εδώ και πολλά χρόνια με ορόσημο το 2015, αλλά δυστυχώ δεν υλοποιήθηκε. Επίση, είναι σημαντική παράληψη στην εκθεσή η απουσία ουσιαστική αναφορά στην ανάγκη να αξιοποιήσει των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην ΑΟΣ ενός κράτους μέλους της Κύπρου δεν αρκεί να αναφέρεται μονάχα δημιουργία ενός μεσογειακού κόμβου φυσικού αερίου είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί στην έκθεση ειδική αναφορά στην ανάγκη να αξιοποιήσει των δυνατοτήτων που δημιουργούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Διότι κάτι τέτοιο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη, ιδιαίτερα στην νότιο και νοτιοανατολική Ευρώπη που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Θεωρώ θετικό το γεγονό ότι αρκετοί συνάδελφοι με τι τροπολογίε του σημείωσαν αυτή τη σημασία των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσογείο. Ε, Επίση, ε, θα, θα πω ότι η αναφορά στην πυρηνική για μα ε, έχουμε διαφορετική άποψη. Εμεί πιστεύω ότι η πυρηνική ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιείται ε, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται για ειρηνικού σκοπού. Έχει τεράστιου ενέχει τεράστιους κινδύνου τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Και έρχομαι σε ένα, το τελευταίο θέμα που το οποίο δεν είναι και του έσχατου. Επειδή αναφέρθηκε και ο κύριο Σόταρκα, ε, θα ήθελα να εκφράσω τη διαφωνία μα στην πρόταση που περιλαμβάνεται στην έκθεση για υποχρεωτική συμμετοχή τη Κομισιόν στι διαπραγματεύσει για διακυβερνητικέ συμφωνίε, καθώ και για αξιολόγηση από την Κομισιόν των συμφωνιών που είναι υποδιαπραγμάτευση. Γνωρίζω ότι αυτό ε, υπάρχει και στο προσχέδιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση. Ε, εμείς θεωρούμε ότι είναι λαθασμένο. Γιατί είναι λαθασμένο. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διασφαλίσει την ενεργειακή τροφοδοσία ή δεν μπορεί να διασφαλίσει την ενεργειακή τροφοδοσία και την επάρκεια όλων των κρατών μελών ούτε έχει πάρει μέτρα για την άρση της απομόνωσης κρατών και υπάρχουν παράδειγμα, να φέρω παράδειγμα τη χώρα μου, η Κύπρος που είναι απομονημένη από τα ενεργειακά δικτύα δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, είναι υποχρεωτική η, συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις και η έγκριση των οποιονδήποτε διακυβερνητικών συμφωνιών. Εμείς θεωρούμε ότι και έχουμε καταθέσει τροπολογία σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να είναι προαιρετική η συμμετοχή της Κομισιόν και να επιβιώνεται μονάχα με σχετικό αίτημα των ενδιαφερμένων κρατών μελών. Μονάχα έτσι δεν θα υπομονωμεύεται η ικανότητα των κρατών μελών να διαπραγματεύονται το περιεχόμενο των συμφωνιών. Και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε καταθέσει πρωτο... Ε, συγκεκριμένες τροπολογίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, thank <clears throat> Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ζητήσω στους συναδέλφους να τηρούν το χρόνο, αν γίνεται, τρία λεπτά για τους σκιώδες. Από τους, ε, για το EFT, ο κύριος Ταμπουρά. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Σαντάργα για τι ε, προσπάθειε που κατέβαλε και για τη συνεργασία που είχαμε. Έχουμε καταβάλει πάρα πολλέ ε, τροπολογίε ε, και νομίζω ότι θα εξεταστούν όλε με πολύ μεγάλη προσοχή. Εμεί είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι πολλά από τα επιχειρήματά μα καλύπτονται και από του άλλου συναδέλφου, στηρίζονται από αυτού. Αναφέρομαι κυρίω στο ότι είναι απαραίτητο να βαδίσουμε προς την ε, ενεργειακή επάρκεια. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει αποκέντρωση και να λαμβάνονται πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Σημαντικό είναι επίσης να έχουμε κατά νου τους ε, στόχους ε, του κλίματος και της ενέργειας, να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να είναι ουσιαστικές οι δεσμεύσεις μας. Πάμε στις μεταφορές εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική μείωση των εκπομπών, να αναθεωρήσουμε την ε, πρακτική εφαρμογή των ενεργειακών μας πολιτικών. Αυτό σημαίνει ότι θέλω να υπογραμμίσω τρία επιχειρήματα, τα οποία κατά την άποψή μας είναι πολύ σημαντικά ο πολίτης θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε ενεργειακής επιλογής. Δεν πρέπει να χάνουμε την κοινωνική διάσταση, όπως επίσης και το ότι είναι απαραίτητο να συμμετέχουν οι πολίτες στην ενεργειακή μετάβαση και εκεί να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν. Δεν μπορεί να υπάρχει μια πολιτική μόνο εκ των άνω προς τα κάτω ε, επιτροπές ε, είναι πάνω από τους πολίτες, θα πρέπει να αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο. Εμείς έχουμε καταθέσει από κοινού με άλλους συναδέλφους τροπολογίες οι οποίες ακολουθούν ακριβώς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω πολλές από τις τροπολογίες να εγκριθούν. Το δεύτερο, ε, θα πρέπει να επιχειρηματολογούμε κάπως ολοκληρωμένα. Η ενέργεια δεν μπορεί να είναι ένα στάσιμο τομέα. Ε, η ενέργεια και η ενεργειακή στρατηγική σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδίδεται σωστή σημασία και εδώ παραθέτω ένα συγκεκριμένο τομέα, ε, σωστή σημασία στην ε, γεωργία. Για κάθε ε, θερμική βαθμίδα ή θερμική νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ισοδύναμο γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε το ενεργειακό μας μείγμα. Τέλος και κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και με όλα τα άλλα είναι ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να λειτουργούν με τη λογική, με βάση τη λογική. Οι αποφάσεις μας δεν θα πρέπει να ε, επιτίθενται στις ε, χώρες προμηθεύτριες γιατί αυτό θα μπορεί να είναι ένα μπούμερανγκ το οποίο θα μετατρέψει την βούληση για ενεργειακή ασφάλεια σε ενέργεια μόνο στη δική μας την Ήπειρο. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος, ε, και προτείνω ε, να μην μιλάτε πάνω από 1,5 λεπτό, γιατί έχω ένα ιδιαίτερα μακροσκελή κατάλογο. Η κυρία Κάλλας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε γιατί πράγματι έχουν κατατεθεί πάρα πολλές ε, τροπολογίες. Αυτό σημαίνει και πάρα πολλή δουλειά. Τώρα, θα ήθελα να σχολιάσω μία σειρά τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Εγώ θα ήθελα να φερθώ στις τροπολογίες εκείνες ε, που δίνουν έτσι μια γενικότερη εικόνα για την προσφορά και τη ζήτηση στην Ευρώπη με στόχο την ε, ενεργειακή ασφάλεια. Ε, αναφέρομαι στο ότι πολλοί λένε οι ενεργειακές μονάδες θα πρέπει να είναι κοντά στον τόπο χρήσης. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα κατά την άποψή μου. Το ίδιο ισχύει και για τις ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να βοηθήσουν τη μετάβαση σε ενέργεια με χαμηλή χρήση άνθρακα, αλλά αυτό στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν μια χώρα ε, ενισχύει ε, τη δική της ενεργειακή παραγωγή και από την άλλη πλευρά των συνόρων υπάρχει ενεργειακή υπάρκεια, αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει διασπάθηση χρήματος. Ε, γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε οι ενεργειακές διασυνδέσεις ε, να διασφαλίζουν το διασυνοριακό εμπόριο και να έχουμε πάντα κατά νου έτσι μια γενική εικόνα και επισκόπηση της ενεργειακής αγοράς. Επίσης θέλω να προβάλλω την ε, ε, υπεραξία της πληροφορίας και της πληροφορικής κυρίως σε σχέση με την ενέργεια. Και κάτι τελευταίο, χαίρομαι που στην ε, έκθεση αναφέρονται, αναφέρεται και το πρόγραμμα διασύνθεσης των χωρών της Βαλτικής. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή τον κύριο Σαντάρκα για την εξαιρετική πραγματικά εργασία που φυσικά αυτή η έκθεση χρήζει και τροποποιήσεων και εγώ θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το ότι σήμερα η Ευρώπη επικεντρώνεται στο στόχο για την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Και υποφέρει πραγματικά σήμερα η Ευρώπη από την ανεπάρκεια, την ενεργειακή και την εξάρτηση τη από χώρε που στο τέλο μπορούν ανα πάσα στιγμή να τη κλείσουν τη στρόφιγγα. Είναι γι' αυτό που λέμε εμεί σήμερα ότι η Ευρώπη δεν έχει πάρα πολλέ επιλογέ αλλά αφού ήδη τη προσφέρεται μια πολύ σημαντική επιλογή διεξόδου για την ευρωπαϊκή στρατηγική και για την ενεργειακή ασφάλεια που είναι η Ανατολική Μεσόγειος που μπορεί να είναι και άλλες περιοχές το τρίγωνο ιδιαίτερα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ φαίνεται ότι είναι πολύ φιλόδοξο, πολύ προσωδοφόρο και με μελλοντική προοπτική. Γιατί να μην εντάξουμε αυτή τη διέξοδο που μα δίνεται για να δείξουμε και εμεί ω Ευρώπη ότι έχουμε εναλλακτικέ λύσει από την προσκόλλησή μα αποκλειστικά και μόνο στη Ρωσία ή σε άλλε αγορέ που στο τέλο αποδεικνύονται αναποτελεσματικέ και ουσιαστικά κρατούν την Ευρώπη νόμιρο. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι για να μπορέσουμε να καταστήσουμε υλοποιήσιμους τους στόχους μας για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να στηρίξουμε χώρες ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την Κύπρο, την Ελλάδα και ευρύτερα την περιοχή με έργα ενεργειακής υποδομής μέσα από το πακέτο Γιούγκερ των 315 δισεκατομμυρίων αλλά και με άλλες πολιτικές για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους μας. Για να μην παραμείνει αυτή η έκθεση ουσιαστικά γράμμα χωρίς περιεχόμενο. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό, θεωρούμε ότι κανένα Ευρωπαίος πολίτη σήμερα δεν μπορεί και δεν πρέπει να στερείται του βασικού κοινωνικού ανθρώπινου αγαθού την πρόσβαση στα θέματα ενέργεια. Και ένα τελευταίο, Επόμενο ομιλητή, κύριε Ζούτσο, και συγγνώμη συνάδελφοι, αλλά πολλέ φορέ είμαι αναγκασμένο σα διακόπτω. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας ε, για αυτή την περιεκτική του έκθεση που καλύπτει όλους τους σημαντικούς τομείς της ενέργειας. Αλλά πρέπει να επιμείνουμε σε δύο θέματα. Το ένα είναι μια πολιτική την οποία ακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό η Ρωσία για να αποκλείσει την Ουκρανία από τη μεταφορά ρωσικού αερίου στην Ευρώπη ξεκίνησε πολύ πριν από την κρίση του 2006 έως 2009 με το North Stream μεταξύ άλλων Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ουκρανία. Η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει μια σταθερή απάντηση σε αυτήν την απειλή έναντι της κεντρικής, ε, ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, προφανώς... Ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα εξακολουθούμε να τις θεωρούμε καθοριστικό πυλώνα της ε, πολιτικής μας για το κλίμα και την ενέργεια. Όμως πρέπει να πράξουμε περισσότερα, να υπάρχει μια ενεργειακή προσέγγιση, προσέγγιση κόστους κόστους-οφέλους και να ε, χρησιμοποιούμε ενδεχομένως και το δυναμικό που προσφέρει κάθε μια περιοχή. Θεωρώ ότι αυτά είναι σημαντικά και πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Ε, προτείνω να κλείσουμε τον κατάλογο. Έχουμε βέβαια άλλους 11 ε, που έχουν ζητήσει ε, να λάβουν το λόγο. Βλέπω δεν διαμαρτύρεται κανείς. Κλείνει λοιπόν ο κατάλογος. Επόμενος ο ο κύριος Κέλλες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση που έχει καταθέσει ο συγητής αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τη σχετική στρατηγική. Αν δεν είχαμε πρόβλημα με την ασφάλεια δεν θα αναφερόταν καν. Και νομίζω το έχουν πει και άλλοι ότι υπάρχει μεγάλη αστάθεια γιατί είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, κυρίως από ασταθή καθεστώτα. Άρα δηλαδή το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε τους δικούς μας τους πόρους και να διαφοροποιήσουμε την τροφοδοσία. Θα πρέπει να αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία στο να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τον αγωγό αερίου που έρχεται από τη Ρωσία. Ε, θα πρέπει ε, να έχουμε μια καλύτερη αγορά στη διάθεσή μας. Αυτό που είπα και προηγουμένως, να αναπτύξουμε τους δικούς μας τους πόρους, κυρίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά να έχουμε περισσότερες διασυνδέσεις ενέργειας ε, γιατί με τον τρόπο αυτό αυτούς τους, τις δυνατότητες διασύνδεσης που υπάρχουν θα τις καταστήσουμε περισσότερες ε, χρήσιμες. Ε, αυτό που λέω δεν είναι ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το ε, σχιστολιτικό αέριο, απλά λέω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε το μείγμα και μάλιστα και με ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Σημασία όμως να αποδώσουμε κυρίως την έρευνα για να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε σε μια σωστή εξέλιξη και Τέλος, όσον αφορά στις μεταφορές, λυπάμαι στην αδελφέλη ο Πρόεδρο, πρέπει να σας διακόψω. Η κυρία Ντάλη, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Θα τα πω τηλεγραφικά γιατί έχουμε μόνο 1,5 λεπτό. Ε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδη εισηγητής διότι ε, ο συμβιβασμός 821 τροπολογιών σίγουρα δεν είναι κάτι αστείο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ε, τονιστεί περισσότερο στην έκθεση κυρίως όσον αφορά το γεγονός ότι είναι απομονωμένα κάποια κρατημέλη, τη διασύνδεση αλλά και τη Μεσόγειο. Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι η επιτάχυνση της εφαρμογής της στρατηγικής υποδομής και σχετικών ε, ε, προγραμμάτων που στόχο έχουν να ε, μειώσουν την απομόνωση των κρατών μελών θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο και θα πρέπει να αναφέρεται υπάρχει και η ε, τροπολογία 628 στην παράγραφο 34. Επίσης, θα έπρεπε να, να επικεντρωθούμε στην επέκταση της διασύνδεσης ε, των δικτύων ε, στις χώρες της Μεσογείου και επίσης θα πρέπει να έχουμε και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή και να έχουμε και καλύτερη ολοκλήρωση των αγορών με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να υπάρχει ασφάλεια φοδιασμού. Τροπολογία 631 είναι όλα αυτά. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και στην 734, η οποία αναφέρεται στα αποθέματα φυσικού αερίου στις χώρες της ε, Βόρειας Αφρικής και τις πρόσφατες ανακαλύψεις που είχαμε στη Μεσόγειο, που θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν και ένα κέντρο για να υπάρχει ένας αγωγός για μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και νέοι αγωγοί με νέα ενεργειακή δυνατότητα που θα αναπτυχθούν στη Μεσόγειο θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ενός δικτύου που θα μπορούσε να συνδέσει τη Βόρεια Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητώ από τον εισηγητή και τους κοιόντες εισηγητής να συμπεριλάβουν και αυτή την παράγραφο στην τελική έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, συγγνώμη που έρχομαι σε τόσο δύσκολη θέση, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, όμως πρέπει να σας διακόπτω. Ο κύριος Εσενίκ. Ετσενίκε. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει θέσει στο προσκήνιο το πρόβλημα της ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, λέει ότι το 2030 ε, το 30% της κατανάλωσης θα είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα έχουμε μειώσει κατά 40% τις εκπομπές αορίου του φαινομένου του θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990. Ο ηγετικός ρόλος ε, στις τεχνολογίες που σχετίζονται με τους στόχους αυτούς ε, είναι ε, καλός και πολλά υποσχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν λοιπόν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, θεωρώ αυτό το οποίο θα ε, το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και δεν κάνουμε είναι το προφανές. Δηλαδή να ζητήσουμε ενεργειακή απόδοση και να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υφή δίκτυα για αυτό το σκοπό. Οι τροπολογίες μας λοιπόν οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, δηλαδή να προχωρήσουμε προς μια σταθερή οικονομία, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει παροχή ενέργειας στους πολίτες μας και θα υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια και κυριαρχία. Κάτι το οποίο, όπως διαπιστώνουμε, έχει μεγάλη σχέση με την πολιτική, διπλωματική και στρατηγική κυριαρχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοραθών Ρουίθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ καταρχάς ε, να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του, όπως και τους κοιόδης εισηγητές. Και επίσης έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες, αρκετές τις έχουν προσυπογράψει αρκετοί συνάδελφοι και θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, ω συμβιβαστικέ τροπολογίε σε αυτόν τον πρώτο γύρο τουλάχιστον συζήτηση. Εμεί θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο των υποδομών και πιο συγκεκριμένα ζητούμε αυτό το οποίο ζητά το Κοινοβούλιο επανειλημμένα όσον αφορά τη διασύνδεση, να είναι δεσμευτικοί οι κανόνες. Επίσης θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις σε χώρες οι οποίες έχουν δυνατότητα να παρέχουν ενέργεια από διαφορεμένες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο από την Ιβυρική Χερσόνησο, που θα μπορούσε να είναι μια πολύ σημαντική πηγή ενέργειας αυτή τη στιγμή. Μια δεύτερη δέσμη τροπολογιών αναφέρεται σε αυτό το οποίο σχολίασαν αρκετοί συνάδελφοι, το να είμαστε πιο φιλόδοξοι προ του στόχου τη απόδοση και τη ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Επίση, όπω είπαν αρκετοί άλλοι συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στην ενεργειακή ένδυα και ζητούμε και ανακοίνωση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να καθορίζει δείκτε για την ανάλυση τη κατάσταση των καταναλωτών και να προτείνει συγκεκριμένε λύσει. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω ο προπολογισμό του ορίζοντα 2020 για την καινοτομία και την έρευνα να ε, αφιερωθεί στην ενέργεια και στην ε, ενεργειακή απόδοση. Ε, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ο Πόλε Ρούμπικ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα είναι το εξής. Νομίζω λοιπόν το θέμα είναι το εξής, ότι όσον αφορά τη μείωση της ε, ενεργειακής ζήτησης, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να περιορίσουμε με τον τρόπο αυτό, τουλάχιστον κατά 20% την ε, ενέργεια από ρηκτά καύσιμα. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε υποκατάστατα με ανανόσιμες πηγές ενέργειας και αυτός ε, είναι και όλος ο στόχος της επάρκειας γιατί η ενεργειακή πολιτική δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την ευρύτερη βιομηχανική πολιτική. Εμείς λοιπόν έχουμε θέσει ως στόχο την βιομηχανική ανασυγκρότηση της Ευρώπης. Ε, έχουμε χάσει το 1,8 της βιομηχανικής παραγωγής. Από το 8 μάλιστα έχουμε χάσει το 2,8 της ε, βιομηχανικής μας παραγωγής. Η βιομηχανία είναι ενεργοβόρος, ε, είναι όμως πολύ σημαντική και αν τελικά από το ΑΕΠ το 30% εκεί αποδίδουμε την βιομηχανική παραγωγή μέχρι το 2030, ε, το να έχουμε σωστό ενεργειακό μείγμα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η βιομηχανικές εγκαταστάσεις να μην φύγουν από την Ευρώπη, να επανέλθουν στην Ευρώπη έτσι ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις απασχόλησης. Αυτός είναι ο βασικότερος στόχος, δηλαδή να έχουμε ε, φτηνή ενέργεια και αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί και η ενεργειακή κατανάλωση. Άρα δηλαδή να έχουμε κατά νου όχι μόνο ότι θα έχουμε εξοικονόμηση, αλλά αν θέλουμε σύγχρονη παραγωγή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η αύξηση της ε, ενεργειακής κατανάλωσης.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 Πρώτον, το θέμα της ε, διασύνδεσης φυσικού αερίου, όχι μόνο ηλεκτρικής ενέργειας. Νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να προσδώσουμε συγκεκριμένη προσοχή. Και δεύτερον, το θέμα της ε, σημαντικής ε, ε, σπουδαιότητες των τεχνολογιών ε, επικοινωνίας και πληροφορικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Να μπορέσουμε να έχουμε ένα ευφιές δίκτυο. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ε, κατάλληλη χρήση και τη συμπεριφορά όλων, όλων των χρηστών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν φραγμοί ε, τεχνολογικής φύσεως ε, στον τομέα των ευφυών δικτύων, ε, οικονομικής φύσεως και ρυθμιστικής φύσεως και θεωρώ ότι εκεί θα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο έγγραφο αυτό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι αξιοσημείωτο. Ο εισηγητής κατάφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Ευχαριστώ. Κύριος Κάρινς και μετά ο κύριος Ποστινάρου θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο σύντομα σχόλια. Άρθρο 40. Ο κύριος Σαουντάργας ε, στην αρχική του έκθεση ε, σε αυτό το άρθρο αναφέρεται στη Ρωσία. Ε, έχει πάνω από 30, αν δεν κάνω λάθο, τροπολογίες επί του άρθρου αυτού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να δηλώσει σαφέστατα πώς έχει κατάσταση. Η Ρωσία είναι ένας ασταθής εταίρος, ε, τώρα το κατά πόσο είναι πολιτικός ε, ασταθής εταίρος ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη εδώ. Δεν συμφωνώ με όλες τις τροπολογίες που κατατέθησαν ε, στο θέμα αυτό. Δεύτερον, το θέμα των διακυβερνητικών συμφωνιών, άρθρο 48. Στο, στην προηγούμενη θητεία ε, συζητούσαμε κατά πόσον ε, ε, θα υπάρχει και προερωτική συμμετοχή αν προσκαλούνται σε αυτές τις διμερείς διαπραγματεύσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας υπενθυμίσω ότι το 90% ζητούσε υποχρεωτική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τα κράτη-μέλη όμως ήταν κατάφορα αντίθετα και στον τελικό συμβιβασμό δεν καταφέραμε να έχουμε υποχρεωτική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρκετοί συνάδελφοι στη συνέχεια συνέχεια δεν υποστήριξαν τον τελικό συμβιβασμό γιατί κατά την άποψή του ήταν πάρα πολύ αποδυναμωμένο. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είναι ευκαιρία να διορθώσουμε το σφάλμα που δεν κατάφερε, αυτό μάλλον που δεν καταφέραμε να επιτύχουμε στην προηγούμενη θητεία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μα υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ ο κύριο Μποστινάρου και ο επόμενο ομιλητή θα είναι ο κύριο Σαφχάουζερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ε, το εξαιρετικό του έργο σήμερα η ενεργειακή ασφάλεια δεν αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού και μόνον, αλλά την ασφάλεια αυτή καθεαυτή ε, λέγοντας, ε, έχοντας κατά νου το γεωστρατηγικό πλαίσιο. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ζητήσω να αναφέρουμε την ε, ανάγκη ε, να συνδυάσουμε την ενεργειακή ασφάλεια με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι τμήμα της συνολικής μας πολιτικής. Δεύτερον, είναι επιτακτική σημασία να υπάρχει συντονισμός με την εξωτερική μας πολιτική, διότι εκεί ακριβώς εφαρμόζονται οι διεθνείς συμφωνίες, όταν αποφασίζουμε την εισαγωγή ή την εξαγωγή ενέργειας. Τρίτον, να μειώσουμε την εξάρτηση από έναν και μόνο προμηθευτή. Ανεξάρτητα από το όνομα του προμηθευτή, αν θα είναι η Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλο. Η εξάρτηση, ο εθισμό σε έναν και μοναδικό προμηθευτή είναι ε, κάτι το οποίο είναι πολύ επιζήμιο. Επίση, θα πρέπει να έχουμε διαπραγματευτική ικανότητα ω Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ο καθένα ε, μεμονωμένα, διότι είμαστε πολύ αποποδεμένοι και πολύ εύκολα μπορεί να μα νικήσει κάποιο όπω η Gazprom. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαφχάουζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν ε, πρόλαβα να καταθέσω τροπολογίες, γι' αυτό θα κάνω κάποιε τεχνικού χαρακτήρα παρατηρήσεις. Όσον αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, εάν θέλαμε να εξοικονομήσουμε 10% από την ενεργειακή μας κατανάλωση, θα έπρεπε τα επόμενα 10 χρόνια να έχουμε ε, επενδύσεις 400 εκατομμύριων ευρώ στον τομέα αυτών της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να μιλάμε. Τρεις ακόμα παρατηρήσεις ουσιαστικές. Η αποτελεσματικότητα είναι αντικείμενο των κρατών μελών με βάση την αρχή της επικουρικότητας και έτσι πρέπει να παραμείνει γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει δεύτερον η, ενεργειακή ε, η προμήθεια ενέργειας βασίζεται σε μακροχρόνια συμβόλαια. 10-20 ετών. Επομένω, οποιαδήποτε πολιτική θα πρέπει να είναι τέτοια μακρά πνοή, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγέ κάθε έναν ή δύο χρόνια. Τρίτον, Ρωσία. Όπω θα σα πούν οι ειδικοί, είναι απαραίτητη για την ε, για το ενεργειακό μείγμα τη Ευρώπη, είναι απαραίτητο πάροχο φυσικού αερίου. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε. Επομένως, αντιθέτως θα πρέπει να τη βοηθήσουμε. Θα πρέπει να βοηθήσουμε μάλλον τα κράτη-μέλη. να συμβάλλουμε έτσι ώστε η Ρωσία να μπορεί με τρόπο πιο ασφαλή να παρέχει την, ενέργεια που μπορεί να παρέχει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επισημάνω τη σημασία της ευρωπαϊκής κοινότητας που συμπεριλαμβάνει χώρες ε, στο, στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Τουρκία, η Σερβία, η Μολδαβία και άλλες Και επίσης σημαντικό ζήτημα είναι οι διαπραγματεύσεις για το TTIP. Το κεφάλαιο για την ε, ενέργεια για την ενεργειακή αποτελεσμα... Ε, ασφάλεια ε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την TTIP. Τώρα, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, μάλλον η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας εξαρτάται από την ενέργεια και τέλος η καθαρή ενέργεια, η χρήση άνθρακα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον είναι και αυτή σημαντική για την ε, ενεργειακή ασφάλεια. Ο κύριος Βαν Στίν από την Κομισιόν, από τη Γενική Διεύθυνση ενέργεια. Θα ήθελα να σας ζητήσω, κύριε συνάδελφε, να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και νομίζω ότι μάλλον δεν θα χρειαστώ ούτε καν τα δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάουνταργας για το έργο του και για την έκθεση και για τον συγκυρασμό των τροπολογιών που ξέρουμε ότι είναι δύσκολη αλλά αξίζει. Δεύτερον, ε, είναι κάτι το οποίο ανέφεραν και πολλά μέλη του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Προφανώς υπάρχει ε, σημαντική μεγάλη σχέση μεταξύ της συζήτησης ε, αυτής της έκθεσης και της ανακοίνωσης της αυριανής της Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση. Αύριο θα έρθει εκπρόσωπος της Επιτροπής για να σας παρουσιάσει το κείμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, να σας ε, ε, πω ότι ήδη αυτά που συζητάμε σήμερα εδώ εμφανίζονται ξεκάθαρα στην ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει η Επιτροπή αύριο. Επομένως θα χρησιμεύσει και ε, η πρωτοβουλία για την Ενεργειακή Ένωση στις συζητήσεις που έχετε για το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την πρόσκληση και πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη διάθεσή σας να σας βοηθήσει όπως επιθυμείτε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ο Σαντάργας, ο συγητής, ε, τα τελευταία δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, για τις ε, παρεμβάσεις τους γιατί για μένα είναι αδύνατον να αναφερθώ σε λεπτομέρειες των παρεμβάσεών σας. Οι παρεμβάσεις αγαπητοί συνάδελφοι ήταν τόσο πλούσιες ε, και μπαίνουν τόσο πολύ σε βάθος ε, στα θέματα που συζητάμε. Θα συνεχίσουμε το απόγευμα με τους και ηγητές. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Να κάνω μόνο δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν, θέλω να πω, έχω την εξής αίσθηση και το λέμε μεγάλη χαρά, βαδίζουμε προς την κατεύθυνση του συμβιβασμού. Αυτή την κατεύθυνση έχουμε ακολουθήσει. Δύσκολο βέβαια αυτό, γιατί έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες, όμως ε, διαφαίνεται ήδη ο στόχος. Από την άλλη, σαφώς και θα υπάρξει διάσταση απόψεων ή άλλες διαφορετικές απόψεις. Αλλά η δουλειά μας είναι να συγκεράσουμε τις απόψεις έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να αποφασίσει επ' αυτών των ε, θεμάτων. Να μπορέσουμε δηλαδή να καταλήξουμε σε συμβασμό, να δούμε ποια θα είναι τελικά η άποψη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και προσβλέπω στη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ ωραία. Η ώρα είναι ακριβώς 10 ε, κλείσαμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ συνάδελφοι και το καταφέραμε αυτό και με ομιλίες ε, του 1,5 λεπτού. Τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα δάση Ψηφίζουμε για τα δάση και για το δασικό τομέα. Ψηφίζουμε. Η συγητής είναι ο Μάρεκ Ιούζεφ Γκρομπάρτσικ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθαν όλα τα μέλη της Επιτροπής. Τέλειο είναι αυτό. Πριν από μία ώρα τα πράγματα δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά από πλευράς παρουσίας των μελών. Προτείνω λοιπόν να μείνετε εδώ κολλημένοι σε αυτή την αίθουσα, εντάξει με κάποιο μικρό διάλειμμα μέχρι τις 6.30 το απόγευμα, γιατί μας έδωσαν την καλύτερη αίθουσα, πολύ ωραία αίθουσα μέσα στο κέντρο του Κοινοβουλίου που θα πρέπει αυτή η αίθουσα να είναι πάντα γεμάτη. Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε. Διαδικαστικό συνάδελφος Εσενίκ, σκιώδης συγητής ε, της ΓΚΟΕ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μου είπαν ότι έχει παρισφρήσει ένα λάθος ε, στην παράγραφο 4, 2. Δεν είναι σωστό ότι την ΚΟΕ έχει υπογράψει αυτό το συγκεκριμένο σημείο στο 4, αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, λέει ο Πρόεδρος, εσείς ως πολιτική ομάδα δεν θέλετε να στηρίξετε τη συμβαστική πρόταση 2, σωστά, σωστά. Άρα δηλαδή την ε, ΚΟΕ την διασβήνουμε, τη σβήνουμε, η ΚΟΕ δεν συμφωνεί με τη συμβαστική πρόταση 2. Καταρχήν, ε, δοκιμαστική ψηφοφορία. Και βάζουμε πάντα στις ε, δοκιμαστικές ψηφορίες την ίδια ερώτηση. Ε, σας αρέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η ερώτηση και πρέπει να ψηφίζετε. Γιατί έτσι γίνεται και μια μικρή δημοσκόπηση για το αν σας αρέσει το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε. Τρεις παραπάνω ψήφισαν στις σοσιαλδημοκράτες, από Τώρα είναι εντάξει, παρακαλώ, εσείς τι θέλετε. Πρόεδρε, η συνάδελφός μου ξέχασε ε, την κάρτα της στο μετρό και πάνε να της την πάρουν. Μήπως ε, μπορούμε να περιμένουμε λίγο. Πρόεδρος, ας ξεκινήσουμε καλύτερα. Υπέρ της τροπολογίας υπαριθμών 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η πέντε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η έξι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η επτά υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 12 υπέρ, κατά, Μισό λεπτό, ηλεκτρονικός έλεγχος, ηλεκτρονική επαλήθευση για αυτήν. Για την 12. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 12 παρακαλώ. Ένας ευρωβουλευτής ε, είναι παραπάνω από ό,τι προβλέπετε από το ΕΛΚ. Από το ΕΛΚ. Πολύ ωραία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αν έχετε καλοσύνη να σηκώνετε ε, καθαρά το χέρι σας, καθαρά ψηλά, γιατί χάνουμε χρόνο. Η 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 30 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 30 ψηφίζουμε ψήφισατε όλοι πάλι περισσεύει ένας από το ΕΛΚ είναι παραπάνω ίσως εγώ λέει ο πρόεδρος Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να είναι ένας παραπάνω. Έκλεισε τώρα η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Υπέρ της 4. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 38 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 40 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για τη 40. Ψηφίζουμε. είναι αρκετοί από το ΕΛΚ που περισσεύουν. Τέλος πάντων, έκλεισε για τις 40, εγκρίνεται. 41, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήτευση για τις 41. Ψηφίσατε όλοι. Ένας από το ΕΛΚ περισσεύει. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 42. Το αποτέλεσμα ήταν 28 υπέρ 28 κατά, σημαίνει απορρίπτεται. Η 42. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 44. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 50 υπέρ κατά εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά νομίζω εγκρίθηκε. Η 53 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Για την 53 ε, ψηφίζουμε. Πάλι περισσεύουν από το ΕΛΚ. Έκλεισε. Ένας περισσεύει. Μισό λεπτό τώρα είναι εντάξει. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Για την 54 όμως, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 54. Δύο περισσεύουν από το ΕΛΚ. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 58 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 58. Ψηφίζουμε. Δυστυχώς ε, περισσεύει ένας από το ΕΛΚ, έκλεισε η ψηφοφορία, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 63 υπέρ, ψηφίζουμε για την 63 παρακαλώ συνάδελφοι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Uh, Δυστυχώς ε, και πάλι περισσεύουν κάποιοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα πολύ καλό. 56 υπέρ 4 ε, κατά. Συνάδελφε, σας συγχαίρουμε. Σας συγχαίρουμε για την έκθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Νομίζω ότι τα καταφέρουμε μια χαρά και από πλευράς χρόνου. Ας πάμε λοιπόν τώρα... Στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και ελπίζω να μείνετε όλοι και για το επόμενο σημείο. No, unfortunately not at all. Δυστυχώς μάλλον κανείς. Because... We must be short here because Oettinger comes. In principle at 30. Uh, dear friends, we've got not more... Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα 20 λεπτό περίπου για το επόμενο σημείο. Επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη, προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση. Θα ήθελα σας παρακαλώ, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, να σας ζητήσω ή να μείνετε εδώ ή σας παρακαλώ αποχωρήστε ησύχως. Δύο πιθανότητες. Είναι αδύνατον, αγαπητοί συνάδελφοι, να συζητάμε εντό τη αίθουσα. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πόχε. Ή ε, φύγετε από την αίθουσα, διότι ε, εμείς θέλουμε με να σας βλέπουμε, αλλά όχι με πηγαδάκια. Ρούμπι. Κύριε Ρούμπιχ, κύριε Ρούμπιχ, παρακαλώ. Είστε μαχνητικό πεδίο, κρατάτε όλους εδώ στην αίθουσα. Λοιπόν, ένα τέταρτο έχουμε για το σημείο αυτό. Πρέπει να οργανωθούμε καλά. Επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη, προώθηση τη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση. Συντάκτη ε, τη γνωμοδότηση, ο συνάδελφο Νεοκλή Ηλικιώτη. Πρόκειται για γνωμοδότηση, επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή είναι Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, ε, ως απάντηση στην έκτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομική, Κοινωνική και Δαφική Συνοχή, επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Πολύ σημαντική έκθεση, συμμετέχουμε και εμείς και θα πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε και να ε, προετοιμάσουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Κύριε Σιλικιώτη, θα ήθελα να σας ζητήσω να λάβετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να, πω, να συμφωνήσω μαζί σας είναι μια σημαντική ε, γνωμοδότηση γιατί η οικονομική κρίση έχει αναντίλεκτα πολύ σοβαρές επιπτώσει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανισότητες και οι διαφορές μεταξύ κρατών μερών αυξάνονται δραματικά όπως και το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, λαών, πολιτών έχει μεγαλώσει επικίνδυνα. Τα μέτρα λιτότητας τα οποία παρουσιάστηκαν ως απάντηση στην, στην κρίση διέλυσαν το βιομηχανικό τομέα, ειδικότερα στον Νότο έχουν οδηγήσει στην αποβιομηχανοποίηση, μείωσαν τις ε, επενδύσεις, απορριθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις, παραβιάζουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και οδήγησαν στο κλείσιμα πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, έχουν χαθεί με την έναρξη της κρίσης πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις, ε, ιδιαίτερα στη μεταπητική βιομηχανία, ανάμεσα στους νέους υπάρχει ένα σοβαρό ποσοστό ανεργία που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια. Ε, απαιτούνται λοιπόν μεταρρυθμίσει και δραστικά μέτρα ώστε να επιτύχουμε και να προωθήσουμε πραγματικά την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα η έφαση θα πρέπει να δοθεί στα κράτη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση καθώς και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης. Ε, είναι σημαντικό να υπάρξει επίση μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιομηχανία. Πρέπει να τονωθεί η πραγματική οικονομία για να μπορέσει έτσι να αντιμετωπιστεί η ανεργία, να προωθηθεί η ανάπτυξη, να δημιουργηθούν νέες θέσει εργασία με ενισχυμένα εργασιακά δικαιώματα και πρόσβαση στη δημόσια υγεία και παιδεία. Ήψιστο στόχο πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η υψηλή ποιότητα ζωής και αξιοπρεπή σε εργασία για όλου. Όσον αφορά τα νέα έργα και τι νέε επενδύσει που προωθούνται με τι χρηματοδοτήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρξει ρήτρα απασχόληση η οποία να ορίζει την υποχρέωση για δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Είναι ε, εξίσου σημαντικό να στηρίξουμε τι δημόσιε επενδύσει οι οποίε θα ανταποκρίνονται στι ανάγκε τη κοινωνία και να δώσουμε ιδιαίτερα κίνητρα στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Για να επιτύχουμε αυτό χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία όπως είναι το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και το πρόγραμμα Κόσμε να προωθήσουμε την κοινοτομία και την έρευνα. Ε, επίσης για να επιτύχουμε πραγματική συνοχή απο, απαιτείται να προωθήσουμε πολιτικές σύγκλησης που να βασίζεται στη διασφάλιση και πρόθεση κάθε χώρα στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και στην προστασία ε, του περιβάλλοντος. Για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι πρέπει να διασφαλίσουμε πως οι πόροι που θα δεθούν αξιοποιούνται χωρίς πατάλες, με πλήρη διαφάνεια κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Πολλά σημεία που έχω αναφέρει συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο που κατάθεσα, αλλά λόγω περιορισμού των λέξεων που έπρεπε να τηρηθεί, ε, θα ε, έχω ετοιμάσει και τροπολογίε. Αναμένω βεβαίω και από του άλλου συναδέλφου να ετοιμάσουν πρωτοπολογίε. Ε, σύντομα θα έχω συνάντηση και με του κοιόδη ηγητή ώστε να συνεργαστούμε για να βγάλουμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα μέσα από αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. Thank you very, very much, Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι, για την παρουσίασή σα. Τώρα έχουμε ε, τους άλλους ομιλητές για ένα λεπτό. Η κυρία Βιρκόνεν εκ μέρους του ΕΛΚ καταρχάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για το έργο του και ευχαριστούμε και για την συνεδρίαση με τους κοιόδης εισηγητές που έχετε προβλέψει. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε εκ νέου διότι δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα χωρίς επενδύσεις και υπάρχουν και τα κονδύλια συνοχής τα οποία οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις κυρίως στο πλαίσιο της στρατηγική 2020 για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Έχουμε την έρευνα, την κοινοτομία, το ψηφιακό θεματολόγιο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν ε, στη χρήση των ε, κονδυλίων να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία, να μπορούμε να εξυγχρονίσουμε την περιφερειακή πολιτική και ταυτόχρονα να φέρουμε στο προσκήνιο την απασχόληση. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος το οποίο συνοδεύει αυτά τα ταμεία, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι ανάλογο και της ε, στήριξης που παρέχεται. Επομένως θα πρέπει να εξετάσουμε την περιφερειακή και τοπική μας πολιτική. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Τάγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, εισηγητή. Συμφωνώ ότι τα Ταμεία Συνοχής είναι όλα ένα και πιο σημαντικά. Ε, τα τελευταία χρόνια ήταν απογοητευτικά. Έχουμε δει αυξανόμενε διαφορέ μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για να μπορέσουμε να έχουμε και πάλι σύγκληση και να βοηθήσουμε τι οικονομίε να εξυγχρονιστούν, αν θέλετε. Θα θέλαμε να τονίσουμε λοιπόν ότι πρέπει να επικεντρώσουμε τις επενδύσεις μας σε θεματικές προτεραιότητες, έρευνα και καινοτομία, ψηφιακό θεματολόγιο, υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οικονομία χαμηλή σε άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα να μεγιστοποιήσουμε τις, ε, την επιρροή που θα έχουμε στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασία. Γιατί αυτά είναι βασικά που μας απασχολούν τα επόμενα χρόνια. Ανάπτυξη και απασχόληση, όχι με λόγια, αλλά με πραγματικές επενδύσεις. Τα ταμεία συνοχή λοιπόν έχουν ε, γίνει πάρα πολύ σημαντικό και ε, θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων μας. Κάθε ευρώ που δαπανώτε θα πρέπει να δαπανάτε με πιο αποτελεσματικό τρόπο και αυτό θα πρέπει να είναι ο κοινό μας στόχος. Ευχαριστώ ο κύριος Τοζανόφσκι εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον εισηγητή και είμαστε κι εμείς βαθύτατα πεπισμένοι ότι ε, θα πρέπει τα κονδύλια αυτά να έχουν μακροπρόθεσμα ε, αποτελέσματα. Θα πρέπει να μην οδηγούν στην ανεργία, θα πρέπει να έχουν ένα χαρακτήρα αποζημίωσης, ε, αποκατάστασης των ελλημάτων αλλά ε, μακροπρόθεσμα. Δεν θα πρέπει με τα ταμεία αυτά να υποκαταθεστούν με τις δυνατότητες ε, ε, που θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τα κάθε κράτες μέλος. Γι' αυτό και ακριβώς χαίρομαι για αυτό το οποίο αναφέρεται στην γνωμοδότηση. Θα πρέπει πραγματικά να υποστηρίξουμε την κατάρτιση, την έρευνα, να υπάρχουν νέα προγράμματα στοιχεία τα οποία θα φέρουν ίσως δευτερογενώς και απασχόληση, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις ε, ε, και να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να δράσουμε και σε κάποιες κοινότητες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαδακα... Μαδραγάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι σε αυτή τη γνωμοδότηση θα, στην οποία πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων, χάρη στο πολύ θετικό έργο του συντάκτη της γνωμοδότησης, θεωρώ ότι υπάρχει ένας κίνδυνος και μια ε, πραγματικότητα. Ο κίνδυνος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να ε, στοχεύει στην έννοια της εγκατάλειψης ε, και στο γεγονός ότι θα πρέπει κατά βάση να ασχοληθούμε με τις ανασότητες και δεν συζητούμε καταλήλως την ευφυή εξειδίκευση, για παράδειγμα, σε περιφερειακούς όρους για να μειώσουμε αυτές τις ανισότητες. Θα πρέπει να επιτύχουμε τέσσερις στόχους και νομίζω ότι αυτοί περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση που θα υποβάλουμε. Ο βασικός στόχος είναι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Όχι απλώς ε, ε, jobs and growth, ω ε, δόγμα που τα τονίζει όλα. Επίσης, ανανέωση τη οικονομία ούτε μικρο ούτε μάκρο, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν μακροπεριφερειακά προγράμματα που θα βοηθούν στην ε, ε, ανταγωνιστικότητα, όχι μόνο στην εμπορική ανταγωνιστικότητα. Τρίτον, ορίζοντας 2020 με την ιδέα της σχετική καινοτομία και αμοιβαία μάθηση σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν κάποια θετικά προγράμματα, πολύ καλά προγράμματα στον τομέα αυτό. Και τέταρτον, η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε αυτά τα προγράμματα της καλύτερης περιφερειακής παραγωγικότητας. Είναι ο καλύτερος κοινός παρανομαστής για αυτή τη διαδικασία της μείωσης των περιφερειακών ισοτήτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρέλ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν, η Επιτροπή μας ε, σε αυτή τη γνωμοδότηση θα πρέπει να αναφέρει κυρίως ε, την σχέση ανάμεσα στα κονδύλια των ε, διερθωτικών ταμείων και το πρόγραμμα Horizon 2020. Να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διασύνδεση από ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο θέλω να καταστήσω απόλυτα σαφές ότι μια γενική ρήτρα για την δημιουργία θέσεων απασχόληση σε όλα τα προγράμματα, μια τέτοια ρήτρα είναι κάτι εκτός πραγματικότητας. Ναι, σημαντικό να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης, αλλά αν τελικά ε, θέλουμε να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση σε σπίτια ιδιωτών. Ε, με τον τρόπο αυτό δεν δημιουργούνται έμεσα θέσει απασχόληση. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο μακροπρόθεσμα και, εν πάση περιπτώσει, όχι με το μέτρο τη αύξηση τη ενεργειακή απόδοση. Εγώ λοιπόν θα ήθελα από αυτού να καταθέσω σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Άλλος κανείς? Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φίλιπ Μόνφορντ, αναλυτής πολιτικής από την ε, Γενική Διεύθυνση Regio. Okay, um, so thank you very much for all these interests. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις ε, για την έκθεση για τη συνοχή. Νομίζω ότι καθόλου λογικές και αιτιολογημένες, ενημερωτικές και σίγουρα υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που άκουσα εδώ τις οποίες ε, θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη ε, για την επόμενη έκθεση κυρίως αυτές οι οποίες ε, σχετίζονται με το στόχο της πολιτικής, την ανάγκη να συνδέσουμε τις δράσεις με την ευρύτερη, ευρωπαϊκή ατζέντα. Αναφερθήκαμε στο Ευρώπη 2020, αλλά υπάρχει και μια συνολική διάσταση. Μόνο αυτό θα ήθελα να σχολιάσω. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ για την άποψή σας επί του ζητήματος και να ζητήσω από τον κύριο ε, Σιλικιώτη να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ σύντομα. Ε, πρώτα πρώτα να πω ότι ε, συμφωνώ και το έθεσε σωστά η κυρία Βρικόνεν από το ΕΛΚΙΑ ε, τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα ε, και ιδιαίτερα τη δυνατότητα πρόσβαση στα προγράμματα ένα πρόβλημα μεγάλο που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να το σημειώσουμε στην έκθεση. Ο κύριο Ντάκα από την ε, S&D νομίζω με μια πρόταση ε, είπε αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος μας ε, όχι μόνο εμά ω Επιτροπή, αλλά συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίοδο κρίση, ανάπτυξη και απασχόληση, όχι μόνο λόγια αλλά και επενδύσει. και είναι σημαντικά μέσα από τι επενδύσει να αναφερθήκαν και άλλοι συναδελφοί και του ευχαριστώ και στου στόχου που πρέπει να τίθενται. Ε, όμως ε, ε, θα πρέπει να πω ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ξεκινούν πρώτα πρώτα από το ίδιο το, το κράτος, από το δημόσιο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να εφαρμόσουμε και πολιτικές για να προσελκύσουμε και ιδιωτικέ επενδύσεις. Και τέλος, να σχολιάσω το θέμα που έθεσε ο, ο κύριος Είναι σημαντικό ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την αργία με προγράμματα κατάρτισης και έρευνα. Ο κ. Μαρακάλ έθεσε του στόχου, νομίζω, που περιλαμβάνονται στην ομοδότηση Και τέλο, αυτό που είπε η κυρία Κρύερα από το ε, είναι σωστό αυτό που λέει, όμω εμεί θέλουμε να σημειώσουμε μέσα από την έκθεση όταν θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσει. Όταν μιλούμε για επενδύσει, πρέπει να υπάρχει και ο στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασία. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που καθίσταται το πρόβλημα της αργίας ιδιαίτερα στους νέους το πιο επίγον, το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνίες ε, της, ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να συνδέσουμε τις επενδύσεις με τη δημιουργία θέσης εργασίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρότασή σας, για τη γνωμοδότηση νομοδότηση της πρωτοβουλίας και τις παρατηρήσεις σας. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για το σχέδιο γνωμοδότησης είναι 26 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι, αυτή την εβδομάδα, 12 η ώρα. Σας παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε την προθεσμία. Με αυτό ολοκληρώνεται το σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα τώρα να σας ενημερίσω ε, για κάποια σημαντικά ζητήματα, αν μου επιτρέπετε. Θα το χωρίσω σε δύο τμήματα. Καταρχάς, ανάθεση εκθέσεων και αποφάσεις ε, που έλαβαν οι συντονιστές. Ανάθεση. Ψηφίσματα και προφορικές ερωτήσεις. Αποφασίστηκε να ε, δώσουμε τις εξής προφορικές ερωτήσεις. Τα big data στην κυρία Κάπελ από τους μη εγγεγραμμένους προφορική ερώτηση με ε, ψήφισμα. Οι συντονιστές αποφάσισαν να αλλάξουν την, να συστήσουν συγγνώμη, την ομάδα επαφής της Acer για να ε, καταρτήσει ε, ένα προφορικό ερώτημα για την έλλειψη πόρων της Acer ε, για την εφαρμογή του Remit. Σχέδιο λοιπόν προφορικής ερώτησης, πολύ σημαντικό ζήτημα και πέραμε τώρα στις αποφάσεις. Οι συντονιστές αποφάσισαν να συστήσουν μια ομάδα εργασίας της ΣΥΤΡΕ για την ψηφιακή Ευρώπη. Όλα τα μέλη της Επιτροπής ΣΥΤΡΕ είναι προσκεκλημένα να συμμετάσχουν ε, και είναι ανοιχτή και σε άλλους, αλλά πρωτίστως αφορά τα μέλη της δικής μας Επιτροπής. Θα αποφασίσουμε στις επόμενες ημέρες για την πρώτη συνεδρίαση, πότε είναι κατάλληλη ημερομηνία για όλους μας, ε, προκειμένου να συνεδριάσουμε και να ξεκινήσουμε έντονες συζητήσεις και εργασίες. Η ομάδα εργασίας λοιπόν ψηφιακή Ευρώπη στην Επιτροπή Ήτρε θα έχει έναν αντίστοιχο ε, τρόπο εργασίας όπως η ομάδα εργασίας ε, για τον ορίζοντα 2020 ε, λίγο πολύ τον ίδιο τύπο θα ακολουθήσουμε. Δεύτερη απόφαση. Αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, Πενσιλβάνια και Ουάσιγκτον. 16 με 20 Μαρτίου. 9 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 16 με 20 Μαρτίου. Αντιπροσωπεία στη Ρήγα και στο Μπάρεκ στην, ε, στον οργανισμό της Ρήγας. 2 με 8 Απριλίου, τρία μέλη από την Επιτροπή Ήτρε και εκτός ποσόστοσης θα είναι ο συνάδελφος Κάρεν, ε, ο οποίος είναι λετονός ε, μέλος της Επιτροπής μας, που εκπροσωπεί και την Προεδρία τρόπον Δεν είδα τον κύριο Έτιγκερ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 Ο Επίτροπος Έτιγκερ λοιπόν είναι και πάλι εδώ μαζί μας. Έξι χρόνια συνεργασίας. Διαφορετικό θέμα αυτή τη φορά, δεν είναι πλέον αρμόδιος για την ενέργεια, αλλά και πάλι σχετίζεται με την ενέργεια. Τα πάντα άλλωστε σχετίζονται με την ενέργεια. Καλώς ορίσατε και πάλι, ε, Επίτροπε Έτιγκερ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε Επίτροπος για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, πολύ σημαντικό ζήτημα για την επόμενη πενταετία και το θέμα είναι ο διαρθρωμένος διάλογος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανταλλαγή απόψεων με τον Γκίντερ Έντιγκερ, Επίτροπο για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, διότι πλέον ε, στην Επιτροπή μας ξεκινούμε το διαρθρωμένο διάλογο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να ε, το εκλάβουμε ως τέτοιο, αφορά και τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων που είναι τόσο σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Επίτροπος Έτιγκερ είναι αρμόδιος για θέματα ε, κρίσιμης σημασίας για την Επιτροπή μας την καλά διασυνδεδεμένη ψηφιακή Ευρώπη, την προστασία δεδομένων, τον κανονισμό για τις τηλεπικοινωνίες, ε, τα πνευματικά δικαιώματα, τα ραδιοκύματα, ραδιοσυχνότητες, μέτρα γι' αυτό, ε, εφαρμογή, εφαρμογή νομοθεσίας ανταγωνισμού και φυσικά θα θέλαμε να υπάρχει και μεγαλύτερη φιλοδοξία στην ε, ε μεταρρύθμιση, για παράδειγμα κανόνες τηλεπικοινωνιών, το ραδιοφάσμα, διαδικτυακή επικοινωνία για πιο ασφαλή δεδομένα και πώς μπορούμε να οργανωθούμε κατά αυτόν τον τρόπο και ε, πολύ ε, ε, σωστές ψηφιακές υποδομές. Φυσικά υπάρχει κοινή αρμοδιότητα με συναδέλφους από άλλες επιτροπές, αλλά πρωτίστως, τα περισσότερα ζητήματα στο, στο χαρτοφυλάκιο του κυρίου Έτιγκερ σχετίζονται με τη δική μας την Επιτροπή, την Επιτροπή Ήτρε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα λοιπόν που ε, είστε εδώ για άλλη μια φορά και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να κάνετε την ε, ε, παρέμβασή σας. Πρόεδρε, αγαπητοί αγαπητέ συνάδελφε Μπούζεκ, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσω μαζί, μαζί σας για τα βασικά θέματα που θέλουμε να δείξουμε το 2015 στον ψηφιακό τομέα. Επίσης, να συζητήσω μαζί σας για διάφορους τομείς και ελπίζω με τον τρόπο αυτό να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο συνάδελφος Αντσίπ ε, τάσεται υπέρ της ε, ολοκλήρωσης ε, της ψηφιακής αγοράς, είναι αρμόδιος γι' αυτό και θέλω να πω ότι η ψηφιακή εσωτερική αγορά είναι ένα θέμα επί του οποίου θα τοποθετηθώ και εγώ. Εμείς λοιπόν φιλοδοξούμε να έχουμε τελικά μια λειτουργούσα ψηφιακή ένωση. Αυτό τον όρο ψηφιακή ένωση τον βρίσκω εξίσου ενδιαφέροντα όπως την ενεργειακή ένωση ή την τραπεζική ένωση ή την ε, κεφαλουχική ένωση. Εμείς λοιπόν επιθυμούμε η ψηφιακή ένωση ε, σημαίνει κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η κοινή, είναι οδηγία για ε, κοινή ψηφιακή αγορά. Στο Ευρωπαϊκό στο Συμβούλιο εχθές ε, συνεδρίασαν ε, διάφορες ομάδες, θα επανέλθουν αυτές, θα ξανασυνεδριάσουν και είμαι αισιόδοξο ότι το Συμβούλιο για αυτή την περίφημη οδηγία NIS ε, για την ψηφιακή ασφάλεια θα αναθέσει εντολή στη λετονική Προεδρία και από πέρυσι από τον Απρίλιο έχουμε βέβαια τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν, λίγο μετά το Πάσχα, νομίζω ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι άμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα ε, στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν θέματα επί των οποίων συμφωνούμε, υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, εγώ είμαι σίγουρος ότι όσον αφορά το θέμα του φάσματος, το Συμβούλιο δεν μπορεί να δώσει καμία εντολή. Αυτό είναι λυπηρό, αλλά το δέχομαι και από την άλλη. Θα προτιμούσα βέβαια αν για την ε, αδειοδότηση συχνοτήτων, εάν για ε, τους πληστηριασμούς ε, για τις ε, συχνότητες δεν θα είχαμε 28 διαφορετικές και κατατμημένες αδειοδοτήσεις γιατί θεωρώ ότι εντωμεταξύ οι συχνότητες είναι πάρα πολύ σημαντικές καθότι έχουμε διασυνοριακούς οικονομικούς χώρους. Άρα δηλαδή θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει συντονισμός των κρατών μελών. Και εφόσον έχουμε εντολή του Συμβουλίου που δεν αφορά όμως το φάσμα, τα αφορά ίσως άλλα θέματα όπως ε, την περιαγωγή και την ουδετερότητα του ε, διαδικτύου. Αυτά πιστεύω θα τα έχουμε και το καλοκαίρι θέλω να ελπίζω ότι θα ξαναζητήσω την εντολή για το ραδιοφάσμα. Το θέμα δεν είναι μόνο τα έσοδα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, αλλά το θέμα είναι το που αφορά αυτά, αφορούν όλα αυτά τον χρήση. Να υπάρχουν λοιπόν καλύτερα αποτελέσματα για τους άμεσα ενδιαφερόμενους, κυρίως για αυτούς που προσφέρουν υπηρεσίες. Όσον αφορά την ουδετερότητα του ε, διαδικτύου, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις διαφόρων κρατών μελών ε, και της Λετωνικής Προεδρίας και θέλω να πω το εξής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ουδετερότητα του διαδικτύου σημαίνει ότι δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει κανενός είδους διακριτική μεταχείριση. Δηλαδή όποιος ενδιαφέρεται για τη ροή δεδομένων ανεξάρτητα με το αν παράγει ή χρησιμοποιεί δεδομένα όλοι αυτοί να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, τόσο σαν αφορά την ποιότητα όσο και το δυναμικό. Τίθεται βέβαια το εξής ερώτημα. Μπορούν να υπάρξουν συγκεκριμένες υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος επί των οποίων όλοι μας ε, επιθυμούμε να υπάρχει μία προνομιούχος μεταχείριση. Παραδείγματο χάρη, αναφέρομαι στο θέμα της οδικής ασφάλειας ε, και της ε, αυτοματοποιημένης οδήγησης. Είχα πάρα πολλές επαφές ε, με κατασκευαστές αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και τους είπα ότι αν τελικά πραγματικά επικρατήσει αυτή η αυτοματοποιημένη οδήγηση χρειαζόμαστε απαραίτητα τη ροή δεδομένων, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει οδική ασφάλεια. Γιατί ας πούμε, ε, ας υποθέσουμε ότι είστε σε μία διασταύρωση στο μέλλον να Έχετε κάποιους από δεξιά, εσείς έχετε βάλει τον αυτόματο πιλότο και σας λέει ο πιλότος, προσέξτε, έρχεται κάποιος από δεξιά, σας το λέω όμως τόσο καθυστερημένα που έχει ήδη γίνει το ατύχημα. Ή άλλη περίπτωση, ε, στον τομέα της υγείας ε, και εκεί υπάρχουν δεδομένα που είναι καθοριστική σημασία. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον εμπορικό τομέα ή αν θέλετε στο θέμα της περιαγωγής. Και εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και θεωρώ ότι η πρόταση της ηλεκτρονικής προεδρίας βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν είναι αρκετά θαραλέα. Βέβαια πρέπει να έχουμε κατά νου, κυρίως την περιαγωγή, ότι δεν έχουν το ίδιο συμφέρον όλοι οι πολίτες, ας πούμε στις χώρες της ε, Μεσογείου ε, και στις χώρες της ε, Βαλτικής τα ενδιαφέροντα αποκλίνουν πλήρως. Δεν μπορεί να υπάρχει λοιπόν το ίδιο κόστος. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια θαραλέα προσέγγιση και θα ξεκινήσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι άλλο, ε, η ενιαία οδηγία, η οδηγία ε, για την ενιαία αγορά αυτή είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και των επικοινωνιών. Γι' αυτό λοιπόν οι υπηρεσίες μου εργάζονται επί του θέματος, ε, χρειαζόμαστε ένα συμπληρωματικό πακέτο, ένα ε, πραγματικά περιεκτικό πακέτο για να υπάρχει μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά τηλεπικοινωνιών. Η σχετική οδηγία είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι αυτού που μπορώ να αποκαλέσω μεταρρύθμιση που πρέπει να υπάρχει κατά τα επόμενα χρόνια στον τομέα της νομοθεσίας. Το copyright και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές στρογγυλές τράπεζες, διοργανώνονται ακροάσεις, ε, υπάρχουν μελέτες, αναλύσεις. Εκείνο το οποίο επιθυμούμε είναι το φθινόπωρο αυτού του έτους να καταθέσουμε μια νομοθετική πρόταση η οποία θα λαμβάνει υπόψη της ε, το πακέτο που υπάρχει για την προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού. Αυτά όλα βέβαια να περάσουν και σε ψηφιακή μορφή. Όσον αφορά το copyright, οφείλουμε να ζητήσουμε μια δίκαιη ισορροπία. Υπάρχουν λοιπόν τρία πράγματα που παίζουν ρόλο ε, σε αυτό το θέμα της ε, προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού. Ε, είμαστε εμείς οι χρήστες, οι πολίτες που ενδιαφερόμαστε, θέλουμε να μορφωθούμε. Ο χρήστης ό,τι ψηφιακό κόσμο θέλει να τα βλέπει, να τα ακούει, να μπορεί να τα διαβάσει. Η επιστήμη και οι βιβλιοθήκες ε, έρχονται και αυτές ε, συμπληρωματικά στον τομέα της μόρφωσης, στην κοινωνία που αναζητά τη μόρφωση. Αυτή είναι η μία πλευρά. Από την άλλη όμως έχουμε τους δημιουργούς. Έχουμε το σεναριογράφο, ε, τον σκηνοθέτη, τον δημοσιογράφο που αναλύει και σχολιάζει, τους μουσικούς έχουμε τους ε, διευθυντές ε, της όπερας, όλους αυτούς οι οποίοι με την πνευματική τους δουλειά και με το ταλέντο τους αυτοί όλοι προσπαθούν και εργάζονται ε, πνευματικά, παρουσιάζουν πνευματικό έργο. Εάν λοιπόν και στο μέλλον θέλουμε να έχουμε πνευματική εργασία, αν δεν θέλουμε μετά από 20 χρόνια να αναφερόμαστε μόνο στον Σέξπιρ, τον Σίλερ και τον Ούντο Γιούργεν, στο Γερμανό, εάν θέλουμε να έχουμε μια γενιά η οποία θα μπορεί και αυτή να δουλέψει στον τομέα ε, της εφημερίδας, του βιβλίου και όσον αφορά την εφημερίδα, δεν εννοώ απαραίτητα το χαρτί, ενώ το περιεχόμενο της ψηφιακής εφημερίδας. Η έρευνα λοιπόν, η ποιοτική παρατήρηση, ο κριτικός αλλά καλός σχολιασμός, η ενημέρωση στην τηλεόραση αν τα θέλουμε όλα αυτά, θα πρέπει εκείνος ο οποίος εργάζεται σε αυτό τον τομέα να έχει και αυτός μία αγορά. Να μπορεί και αυτός να έχει κάποια έσοδα, γιατί αλλιώς προφανώς και δεν θα ασχοληθεί με αυτά τα επαγγέλματα. Και υπάρχει και ενδιάμεσα ένας άλλος χώρος, ο ενδιάμεσος χώρος είναι οι εκδότες, ή ε, τα τηλεοπτικά κανάλια, είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτικά πρόσωπα δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου, έχουμε τους παρόχους, έχουμε τις πλατφόρμες, έχουμε όλους αυτούς τους ενδιάμεσους που ασχολούνται με τη μεταφορά, με το εμπόριο αλλά και με την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων. Εκείνο λοιπόν το οποίο είναι σαφές είναι το εξής. Εφόσον ε, μιλάμε και θέλουμε αυτή την ψηφιακή αγορά, αμφισβητείται η αρχή της ε, εδαφικό, της περιφερειακής, της εντοπιότητας μάλλον. Αμφισβητείται η αρχή της εντοπιότητας. Δηλαδή, θα πρέπει πλέον να έχουμε μία και μόνο περιφέρεια. Εγώ τάσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ αυτής της αρχής. Όχι διαφορετικές ε, ε, περιφέρειες, ε, ένα κατακαιρματισμό της περιφέρειας. Εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρχει η εθνική πρόθεση κινηματογραφικών ταινιών. Παραδείγματο χάνει στην Αυστρία, όταν πωλείται και προωθείται μία ταινία, αυτό θα μπορεί να σημαίνει ότι αυτή ε, μπορεί να προσφερθεί χωρίς κόστος ε, και στις άλλες χώρες, ε, στον Ρωμανό Βασίλειο ή οπουδήποτε λούπ. Βεβαίως με παράλληλη εισπραξή εσόδων. Άρα καταλαβαίνετε, αυτή η ισορροπία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Εμείς ευελπιστούμε. ότι η οδηγία, η περίφημη οδηγία ΝΙΣ, η οποία αφορά την κυβερνοασφάλεια, αυτή η οδηγία ε, θα εγκριθεί και μάλιστα πριν από το καλοκαίρι. Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας δεδομένων, αυτό το θέμα είναι υψίστης σημασίας, γιατί ειδικά τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε γεγονότα τα οποία καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι τα συστήματα με τα οποία αποθηκεύουμε, μεταφέρουμε και προσφέρουμε δεδομένα, αυτά τα συστήματα είναι πολύ ευάλωτα, είναι εκτεθειμένα, έρμεα θα έλεγα, όλων κάθε μορφής επίθεσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, η η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ο χρήστης και αυτός έχει προχωρήσει πάρα πολύ και δυστυχώς υπολείπεται η ασφάλεια των δεδομένων. Εάν λοιπόν δεν θέλουμε να τα μόνο με την ασφάλεια των δεδομένων, θα πρέπει να συνδυάσουμε την ασφάλεια των δεδομένων και με την χρήση των δεδομένων. Γιατί τελειώ υπάρχει και να καταστραφούν τα πάντα. Γιατί αν ισχύει ότι ο κατασκευαστής των καρτών SIM, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτών των καρτών, δεν μπορεί να μας προσφέρει την ασφάλεια των κινητών τηλεφώνων εάν ισχύει ότι έξω από την Ευρώπη, από τη Ρωσία, από τις ΗΠΑ, από την Κίνα, από οπουδήποτε υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να εξαπολυθούν στην ευρωπαϊκή ασφάλεια δεδομένων, καταλαβαίνετε αυτό είναι πρόβλημα και για τον πολίτη, αλλά πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ενεργειακές υποδομές, για τις μεταφορικές υποδομές και κατόπιν τούτου για τη δημόσια ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όλα αυτά ελοχεύουν κινδύνους για τη βιομηχανία μας, για την οικονομία μας, γιατί αυτό που παλαιότερα ήταν η οικονομική κατασκοπία, όπου οι κατάσκοποι πήγαν επιτόπου στα εργοστάσια και εκεί έπαιρναν φωτογραφίες, έκαναν φωτοαντίγραφα, εκεί έκαναν σχέδια, κατάσκοποι και κλέβανε, εν πάση περιπτώσει, διάφορα σχέδια. Σήμερα η οικονομική κατασκοπία γίνεται ψηφιακά. Ε, μπορεί κανείς να παρακολουθεί ψηφιακά το τι γίνεται στην Γουατεμάλα, στη Μόσχα, οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε να κάνουμε με ένα ε, καθοριστική σημασία θέμα και σχετικά με την έδρα που θα έχουν ε, οι βιομηχανικές μονάδες στην Ευρώπη. Να είναι δηλαδή προστατευμένες από ψηφιακές επιθέσει. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και οι χρήστες, σας είπα, υπολείπεται η ασφάλεια των δεδομένων τουλάχιστον κατά 10 έτη. Ε, μετά την θέσπιση της οδηγίας νη για την κυβερνοασφάλεια, σας ανακοινώνω ότι θα υπάρχουν και άλλα μέτρα ε, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη χρήση των δεδομένων από την ασφάλεια των δεδομένων. Και φτάνω τώρα στο προτελευταίο σημείο της παρέμβασης μου, κύριε Πρόεδρε, το REFIT για ε, την οδηγία περί οπτικοακουστικών μέτρων. Ε, θα την ολοκληρώσουμε και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ελέγξει ε, το ε, ποιες παράγραφοι και ποια άρθρα είναι πλέον πεπερασμένα ή είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Και αφού το κάνουμε αυτό θα προβούμε σε αναθεώρηση. Δηλαδή, ο εξυγχρονισμός ο, η, ισοπαίδωση της οδηγίας που προέρχεται από το 2007 αυτή ισχύει, έχει ξεπεραστεί αυτή η οδηγία. Άρα δηλαδή το αργότερο μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους θα πρέπει να έχουν κατατεθεί νέες προτάσεις. Τελευταία μου παρατήρηση, υποδομές. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, μπορέσαμε να σας παρουσιάσουμε ε, την, το πρόγραμμα του κύριου Γιούγκερ. Ε, μας ήταν ενθάρρυνση αυτό για μας, γιατί νομίζουμε ότι μπορούμε να αποχωρήσουμε στον θέμα, στον τομέα του ψηφιακού κόσμου. Η ψηφιακή ένωση μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον υπάρχει μια αποτελεσματική ψηφιακή υποδομή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ήρθαμε σε επαφή με τις τηλεπικοινωνίες της Ευρώπης, με τον χρηματοπιστωτικό κόσμο της Ευρώπης, με την ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης, οργανώσαμε στρογγυλές τράπεζες και συζητήσαμε διαμακρών το ποια είναι η απαραίτητη βάση συγχρηματοδότησης ή πώς πρέπει να συρρυκνωθούν οι κίνδυνοι έτσι ώστε να μπορούμε ταχύτερα να περάσουμε σε ένα δίκτυο ε, το οποίο να καλύπτει ακόμα και τις ε, απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. better. Για αυτή την παρέμβαση, για αυτό το σημαντικό θέμα, όπως είπατε, που πρέπει να ρυθμιστεί. για το ζήτημα της ψηφιακής Ευρώπης, τι λέμε. Συμφωνούμε ότι η καλύτερη λύση είναι εκείνη που θα βρεθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στον κράτον μελών. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ έχουμε διαφορετική εξελόγηση της αρχής της επικουρικότητας. Εάν η απάντηση είναι ναι, τότε θα πρέπει να προετοιμαστεί ένα νέο πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες γιατί φαίνεται λοιπόν ότι το καλύτερο ε, επίπεδο στο οποίο μπορεί να λυθούν τα προβλήματα της ψηφιακής Ευρώπης είναι εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονιστές, ο κύριος Κάριντς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε την Τραπεζική Ένωση, την Ενεργειακή Ένωση, την Ψηφιακή Ένωση φαίνεται όλες αυτές οι ενώσει συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε κανείς να πει. Αστείευαμε. Για το ζήτημα τη ουδετερότητας των δικτύων. Φυσικά ο στόχο εδώ είναι να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση, αλλά υπάρχει και το ζήτημα της να μπορεί να θέτει κανείς προτεραιότητες, για παράδειγμα, ε, και εξηγούμε. Για τα δεδομένα που αφορούν στον τομέα τη υγεία ή της, ε, τον αυτόματο πιλότο σε αυτοκίνητα. Δεν είναι τραγικό να χρειαστεί να περιμένει κανείς ένα-δύο δευτερόλεπτα εάν τα δεδομένα που μεταφέρονται, τα δεδομένα που τον αφορούν είναι τα δεδομένα μιας ηλεκτρονικής αγοράς, αλλά εάν μιλάμε για τα δεδομένα οδήγησης, εκεί χρειάζεται, είναι απαραίτητο να μην υπάρχει μια καθυστέρηση. Επομένως λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση και άρα την ίδια ταχύτητα για την ίδια τιμή, αλλά αυτό θα οδηγούσε στους στην κατάσταση οι καταναλωτές εκείνοι που να μην έχουν ανάγκη αυτό το ευρωζώνη σε αυτή την ταχύτητα να πληρώνουν περισσότερο για ένα αγαθό που δεν χρειάζονται. Μια άλλη ερώτηση, γιατί στο παρελθόν το Κοινοβούλιο έχει γκρίνει ένα ψήφισμα για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Και αυτό ο τύπος το παρουσίασε ως επίθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά της Google. Και αν δεν απατώμε, ο Ομπάμα πρόσφατα είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο να προστατεύσει την δική της αγορά παρά να εμπλακεί σε ανταγωνισμό με τις υπόλοιπους παίχτες. Και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη της Επιτροπής με ποιο τρόπο μπορεί να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι ε, εταιριών και φορέων οι οποίοι προσπαθούν να επιδιώξουν οικονομικό όφελος. Ο κύριος Νίκα, εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση και χαιρετίζω την πρόθεσή σας να εργαστείτε στον τομέα της στρατηγικής για την ψηφιακή ολοκλήρωση και της τηλεπικοινωνίας στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε τώρα, μετά την ε, παρουσία σας εδώ, ποιος ακριβώ είναι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τα θέματα αυτά στην Επιτροπή. Έχω τέσσερα ερωτήματα να σας θέσω. Πράγματι, δεν είναι δυνατό να υπάρξει μια ενιαία ψηφιακή αγορά εάν υπάρχει κατακαιρματισμός 28 διαφορετικές αγορές στα κράτη-μέλη. Πρέπει να φροντίζουμε η πρόσβαση στα δεδομένα για τους πολίτες να είναι ανοιχτή οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτοί και χωρίς οικονομικό κόστος ε, υπερβολικό. Ε, συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα με το πολύ μεγάλο κόστος της περιαγωγής. Θα πρέπει επίσης να μην ξεχνούμε ότι Ορισμένες υπηρεσίες, όπως εκείνες που πρέπει να ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες, πρέπει να έχουν μια πιο γρήγορη πρόσβαση ε, στο ίντερνετ, στις επικοινωνίες. Για το ζήτημα του, της χάρτη, του χάρτη των συχνοτήτων, πρέπει να ξεπεράσουμε τα εθνικά εμπόδια και νομίζω ότι αυτός ο κατακαιρματισμός στο εθνικό επίπεδο όσον αφορά στην κατανομή των συχνοτήτων είναι ένας από τους λόγους που βρισκόμαστε πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ. Γιατί οι πάροχοι προσπαθούν να δημιουργήσουν από την πλευρά τους νέα δίκτυα και να παράσχουν νέου τύπου υπηρεσίες. Το 4G και άλλες. Αλλά η Ένωση δεν τους δίνει τα κίνητρα που θα χρειάζονται και δεν τους δυσκολύνει σε αυτή την προσπάθεια. Και κάτι ακόμα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, Θα πρέπει να εργαστούμε στον τομέα αυτό και κυρίως στον τομέα της πιστοποίησης για να αυξηθεί ε, η, εμπιστοσύνη των πολιτών στα ηλεκτρονικά συστήματα αγοράς, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες γενικότερα. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα λοιπόν για την πιστοποίηση, για την έκδοση ε, πιστοποιητικών ασφάλειας. Αυτά την πλευρά. Ευχαριστώ. Μέρος του ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα κύριε Επιτρόπε. Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη συζήτηση για αυτά τα θέματα με εσάς. Είναι πολλά τα θέματα που ανοίξατε και η σημερινή συνάντηση είναι μια, ένα πρώτο βήμα για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα ε, της ψηφιακής στρατηγικής, των δικτύων κτλ. Ε, είναι τα θέματα αυτά εξαιρετικά ε, βρέως χαρακτήρα, είναι ένας τομέας ο οποίος κινείται γρήγορα, αλλάζουν τα πράγματα γρήγορα, υιοθετούνται νέα πρότυπα πολύ γρήγορα και νέες υπηρεσίες εμφανίζονται. Το οποίο μας οδηγεί στην εξής φιλοσοφική ερώτηση. Τι νόημα έχει και μέχρι πού πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίζει κανόνες στον τομέα αυτό. Μήπως η παρέμβαση των κρατών και της Ένωσης γενικότερα στην πραγματικότητα είναι μια τροχοπέδη για την τεχνολογική ανάπτυξη και μήπως τελικά δημιουργεί επιπλέον προβλήματα τα οποία εκ των υστέρων προβλήματα που ίδια δημιούργησε θα προσπαθήσει να λύσει. Μήπως λοιπόν υπάρχει υπερβολική ρύθμιση του τομέα αυτού. Έχει νόημα το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχουμε ήδη εγκρίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μήπως καλύτερα να εξετάσουμε ποια στοιχεία αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου έχουν ήδη ξεπεραστεί από την αγορά και μετά να δούμε με ποια νέα φιλοσοφία μπορούμε να προστατεύσουμε αυτή την αγορά, να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γιατί διαπιστώνουμε αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από την τεχνολογία. Αν κάποια στιγμή καταστρεφόταν η πρόσβαση στο ίντερνετ ή στα δίκτυα θα είχαμε αμέσως ε, προβλήματα σε όλα τα άλλα συστήματα, τα ενεργειακά, το τραπεζικό κτλ. Θέτω λοιπόν το εξή ερώτημα. Βοηθάει η σημερινή νομοθεσία ή μήπως πρέπει να την αντικαταστήσουμε για την Άλντε. Εάν θέλουμε το ίντερνετ να συνεχίσει να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να συνεχίσει να παραμένει ανοιχτό. Όσο πιο δύσκολη γίνεται η πρόσβαση στο startup στο ίντερνετ, τόσο μικρότερες δυνατότητες υπάρχουν και καινοτομία. Τόσο λιγότερες δυνατότητες υπάρχουν και καινοτομία. Αναφερθήκατε σε εξαιρέσεις που θα μπορούσαν να γίνονται στην ε, δημόσια προμήθεια ε, ψηφιακών υπηρεσιών, υπηρεσιών δικτύου και αναφερθήκατε πιο συγκεκριμένα στις επικοινωνίες για τα έξυπνα οχήματα. Να καταλάβω γιατί χρειάζεται αυτή η εξαίρεση σε ένα συγκεκριμένο τομέα σήμερα, αλλά τι θα γίνει στο μέλλον, εάν αρχίσουμε να κάνουμε τέτοιες εξαιρέσεις, θα, θα μπορούσαν τα μεγάλα μονοπόλια να αξιοποιήσουν τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά και με το παραθυράκι των εξαιρέσεων στην πραγματικότητα να δημιουργήσουν μολευκές καταστάσεις. Με ποια φιλοσοφία λοιπόν θα μπορούσαμε να δεχτούμε εξαιρέσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν χρειάζονται, δεν, δεν, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Όσον αφορά την φορολόγηση και την επιβολή τελών στη χρήση του ίντερνετ. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε, ε, έχουμε διαπιστώσει σε κάποιες χώρες, σε κάποια κρατημέλη συγκεκριμένα. Στη Γαλλία και άλλες ότι είναι ένα σύστημα, ένας μια πολιτική που χρησιμοποιείται για να περιορίσει την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν ξεκινήσουμε όμως τέτοιες διαδικασίες, όχι απλώς θα κατακαιρματιστεί το ίντερνετ, όχι απλώς θα, δημιουργήσουμε εμπόδια στις επικοινωνίες, αλλά αυτό θα μας απομονώσει κιόλα. Τέλος, σε αναφορά την ψηφιακή, ψηφιακή επιχειρηματικότητα και πώς μπορούν να εισαχθούν περισσότερο οι νέες τεχνολογίες γενικότερα στις βιομηχανίες, στην, στην ε, στην οικονομία. Θα ήθελα να μου πείτε τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε στον τομέα αυτό. Κύριος Χέρτς, για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Έρτς. Τρεις ερωτήσεις. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Επίτροπε, είστε υπέρ της ε, μερικής ε, αναστολής της ουδετερότητας του δικτύου. Τα επόμενα χρόνια θα κάνετε ακριβώς αυτό, καλά κατάλαβα. Θα μπορούσατε να μου διευκρινίσετε κατά πόσον ε, αντελείβει σωστά. Αν αυτό σκοπεύετε να κάνετε, θα ήθελα να το διευκρινίσετε. Αυτό θα μπορούσε να αφορά διάφορες ε, υπηρεσίες και θα μπορούσε ίσως να δικαιολογήσει και κάποιες πολιτικές ε, για να υπάρχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τραπεζικές υπηρεσίες, κατεπίγουσα ε, βοήθεια. Ε, τι ακριβώς όμως θα σημαίνει αυτή η μερική αναστολή του ισοδετερότητας του δικτύου. Δεύτερον, ε, δικαιώματα δημιουργών και πράσπιση του copyright. Θα ήθελα να ξέρω κάποια περισσότερα πράγματα. Τι ακριβώς θα γίνει το 2015, πιο συγκεκριμένα, ποια στάδια θα υλοποιηθούν, με ποιον θα δράσετε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι ακριβώς θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε λίγο τις προθέσεις σα. Και τρίτη παρατήρηση, ε, η προστασία των δεδομένων. Ε, θα διαβάζετε φυσικά τον τύπο, όπως και εγώ. Ε, υπήρξαν σημαντικά φαινόμενα hacking, εμπιστευτικότητα των δεδομένων και φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον καμία ασφάλεια στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτός ο προστατευτισμός ε, της ε, προστασίας των ε, προσωπικών δεδομένων είναι κάτι το οποίο φυσικά επιθυμούμε όλοι. Είμαστε όλοι υπέρ της προστασίας των δεδομένων. Αλλά όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων τι συνεργασία υπάρχει με τους άλλους επιτρόπους, τον Επίτροπο Τίμερμανς ή οποιονδήποτε άλλον είναι αρμόδιος. Πώς θα διαρθρωθεί αυτή η συνεργασία. Διότι οτιδήποτε θα κάνετε σε επίπεδο ψηφιακού θεμετολογίου ε, είναι ε, κάτι το οποίο παρακολουθεί και η Σύμβαση του Άρχους αλλά και άλλοι. Η προστασία των δεδομένων των πολιτών δεν είναι εγγυημένη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ από το EFTD ο κύριος Μπορέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροβε, όσον αφορά το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Απρίλιο πέρσι ένα σαφή ορισμό και αρκετά ευρύ του τι ακριβώς εννοούμε με την έννοια ουδετερότητα του δικτύου. Επομένως, το πολιτικό όραμα αυτού του κοινοβουλίου είναι εκπεφρασμένο και νομίζω σαφέστατα εκπεφρασμένο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, επί παραδείγματι, έχουν μια πολύ στεναρή και σαφή στάση υπέρ της ουδετερότητας του δικτύου. Πολύ σύντομα. Μήπως θεωρείτε ότι η απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ ε, δεν θα έπρεπε να είναι και ένα κίνητρο για την καινοτομία. Ε, πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάπελ από τους μία γεγραμμένους. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε και Πρόεδρε. Ε, όσον αφορά αυτά που είπατε για την ψηφιακή ένωση, σήμερα το πρωί συζητήσαμε για το θέμα αυτό και με τον Επίτροπο που συζητάγαμε για την κεφαλουχική Ένωση. Το ψηφιακό θεματολόγιο είναι πολύ σημαντικό. Η ενίσχυση μορφών χρηματοδότησης, κυρίως για επιχειρήσεις που ασχολούνται με δεδομένα, να υπάρχουν εναλλακτικέ δυνατότητες χρηματοδότησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ψηφιακό τομέα μας ε, μιλήσατε για τις προτεραιότητές σας για το 2015. Η οδηγία NIS είναι πολύ σημαντική. Μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων όπως και μεταρρύθμιση του copyright. Πολύ σημαντικά αυτά. Αυτό όμως που δεν άκουσα, ίσως πρέπει να το τονίσετε και γι' αυτό ρωτάω, είναι η σύγκριση Ηνωμένε Πολιτείε και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουμε πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις που ασχολούνται με δεδομένα και η Ευρώπη υπολείπεται. Ε, Επίσης, πολλές φορές αναφέρεται ότι ο στόχος σας είναι να γίνουμε παγκόσμιοι παίκτες ή να υπάρχουν πολλοί παγκόσμιοι παίκτες στην Ευρώπη. Ε, και αυτό είναι σημαντικό γιατί βλέπετε ότι τώρα ε, υστερούμε όσον αφορά τη βιομηχανική απόδοση. Και επίσης οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι ασυντόνιστες. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχουν επιτυχημένες εταιρείε δεδομένων. Είπατε ότι θα υπάρχουν προγράμματα φάρος, εμβληματικά προγράμματα που αναφέρονται και σας ερωτώ ε, τι θα γίνει τώρα με αυτά τα εμβληματικά προγράμματα και πώς ακριβώς ε, θα πλησιάσετε το στόχο να γίνουμε ε, παγκόσμιοι παίκτες στο θέμα του ψηφιακού θεματολογίου. Σας ευχαριστώ. Verehrte Damen und Herren Abgeordnete, zu Ihren Stichworten einige konkrete äh, Antworten, aber vorausgeschickt Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω το εξή. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι το εξή. Ο ψηφιακό κόσμος ε, έχει μια τελείως διαφορετική ταχύτητα αλλαγή. Δηλαδή, ο ψηφιακό κόσμος αλλάζει πάντα γρηγορότερα. Και εκεί όπου βάζουμε προδιαγραφέ ή νομοθετούμε ή ρυθμίζουμε, σε αυτού του τομεί είμαστε πάρα πολύ αργοί. Για σκεφτείτε λιγάκι μία οδηγία στον ψηφιακό τομέα. Είτε είναι λευκή βίβλος, είτε πράσινη βίβλος, είτε ανακοίνωση, είτε πρόταση νομοθετήματος. Πρέπει να περάσει ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς τα κάνετε γρήγορα. Μετά το Συμβούλιο για ένα χρόνο δεν κάνει τίποτα. Ο βασικός κανονισμός ε, για την προστασία εντομένων ήταν μπλοκαρισμένος ε, στο Συμβούλιο για ένα χρόνο. Όσον αφορά την οδηγία 1S, τον Απρίλιο εσείς τοποθετηθήκατε πολύ σωστά και το νωρίτερο το Μάρτιο θα έχουμε την εντολή. Δηλαδή χάσαμε ένα χρόνο. Μετά όλα αυτά θα πάνε στον ε, τριμερή διάλογο. Μέχρι το τέλος του έτους ελπίζουμε να εγκριθεί μετά η εφαρμογή στα κρατημέλη, μετά τα εθνικά νομοθετήματα από μία ή δύο βουλές. Δηλαδή χρειαζόμαστε τέσσερα χρόνια. Και σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, αυτά που πρότεινε η Κομισιόν πριν από τέσσερα χρόνια δεν είναι πια επίκαιρα, είναι ξεπερασμένα. Γι' αυτό λοιπόν θέτω το εξής ερώτημα προς όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Μπορούν να υπάρχουν τομείς όπου τα τέσσερα χρόνια ή και τα τρία δεν είναι πρόβλημα. Σε άλλους όμως, ε, σε άλλους τομείς, εάν στον ψηφιακό τομέα, κυρίως στην ανταγωνιστικότητα για την Νότια Κορέα, την Κίνα και την Ιαπωνία. Με τη δική μας την πολιτική, με τις δικές μας τις ρυθμίσεις θέλουμε να θέσουμε παγκόσμιους κανονισμούς και θέλουμε να έχουμε κύρος στον κόσμο και εάν οι νέοι πρέπει να δεχτούν τις δικές μας προτάσεις για το διαδίκτυο, τότε καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να έχουμε ένα σωστό ρυθμό, μια σωστή ταχύτητα. Γι' αυτό λοιπόν την όλη διαδικασία του να αποφασίζουμε στον τομέα τον ψηφιακό, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Και θα επανέλθω. Δηλαδή τι σημαίνει, σημαίνει μικρότερες διορίες, να σκεφτόμαστε περισσότερο, να δουλεύουμε ουσιαστικότερα και να αποφασίζουμε γρηγορότερα. Γιατί αλλιώς που δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το ρυθμό αυτού που απαιτεί η ψηφιακή τεχνολογία. Πριν από 7 χρόνια δεν υπήρχαν τα iPhone και μέσα σε 7 χρόνια υπάρχουν οι κανονισμοί εκείνοι οι οποίοι είχαν εγκριθεί από την Κομισιόν πριν από 7 χρόνια. Δουλεύουμε με ρυθμούς του Νεάντερταλ. Και αυτό το λέω και ως αυτοκριτική προς εμένα, προς τις υπηρεσίες μου, προς όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τελείως διαφορετικές ρυθμίσεις για την ψηφιακή νομοθεσία. Δεύτερον, γιατί χρειαζόμαστε τις ρυθμίσεις. Τις χρειαζόμαστε διότι η ψηφιακή οικονομία τίνει προς τα μονοπόλια. Όποιος λοιπόν ανακαλύψει σήμερα μία πλατφόρμα ή αναπτύξει ένα λογισμικό ή όποιος είναι ηγέτης της αγοράς, ακόμα και αν είναι κρατική επιχείρηση, αυτός έχει πάντα τη δυνατότητα να κυριαρχήσει στην αγορά ή να δημιουργήσει μονοπόλιο. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ρυθμίσεις έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός, έτσι ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των χρηστών. Άρα δηλαδή ειδικά στον ψηφιακό κόσμο χρειαζόμαστε μια έξυπνη νομοθέτηση ευφύης, ρυθμίσεις πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλους τομείς της ε, οικονομίας μας και της κοινωνίας μας. Όσον αφορά το copyright, θέλουμε πολύ συγκεκριμένα το φθινόπωρο αυτού του έτους να καταθέσουμε μία δέσμη νομοθετημάτων όπου θα τίθενται σημαντικά θέματα του ε, δικαίου περί δικαιωμάτων δημιουργού αλλά αυτά ε, κυρίως για τον ψηφιακό κόσμο και θέλουμε να επιφέρουμε την ισορροπία ανάμεσα στο διαδίκτυο αφενός και στην πνευματική εργασία αφετέρου. Εκεί λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε και το εξής ερώτημα. Οι ε, εκδότες, οι εφημερίδες, εκδότες εφημερίδων μας είναι σημαντικοί. Η ραδιοφωνική σταθμή, η τηλεοπτική σταθμή μα είναι σημαντική, γιατί στον ψηφιακό κόσμο φαίνεται όλο και περισσότερο ότι ο χρήστης πάει κατευθείαν στο αντικείμενο και δεν χρειάζεται τον ενδιάμεσο. Έτσι λοιπόν είδατε τι έγινε με την εταιρεία Uber στα ταξί ή το, τις αγορές online σε σχέση με την ένδυση ή με τα βιβλία πάλι, η Amazon που δίνει απευθείας τα βιβλία. Τι σημαίνουν αυτά, ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ε, νομοθεσία περί ψηφιακού ε, copyright. Αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ρυθμισμένη διάδοση στην αγορά το έργο να μπορεί κανείς να το αποκτήσει σε προσιτή τιμή, ε, γρήγορα και χωρίς ε, διακρίσεις. Σήμερα θα, γίνει μια, θα λάβει χώρα μια συνέντευξη τύπου και σε αυτήν θα ε, υπάρξουν διευκρινήσεις για αυτά που γίνονται στην αγορά. Δώστε μας λοιπόν χρόνο μέχρι σήμερα το βράδυ. Δεν πρέπει να δουλεύουμε με προκαταλήψεις, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι αυτά τα οποία άκουσε κανείς για το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να τα εκλαμβάνει ως ε, απόψεις, οι οποίες όμως δεν αφορούν και δεν επιτίθενται στα κινητά τηλέφωνα. Στα κινητά τηλέφωνα υπάρχει και η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και της επιχειρηματικής σφαίρας. Να μην είναι δυνατόν να υπάρχουν επιθέσεις από hackers. Προφανώς αυτά ισχύουν και για τις μυστικές υπηρεσίες ε, ε, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα τύγει και αφορά το Horizon 2020. Στον προϋπολογισμό μας ε, για την ε, έρευνα ε, προβλέπεται η συγχρηματοδότηση προγραμμάτων στον ψηφιακό κόσμο. Ένα δίστο χρόνο, αυτό είναι το ποσό που έχουμε προβλέψει. Και το θέμα είναι τα κονδύλια αυτά να μην διατίθενται μόνο στη βιομηχανία, αλλά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε νεοφυείς επιχειρήσεις, τα startups. Άρα δηλαδή με ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να στηριχθούν οι νέες ιδέες, τα νέα προϊόντα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητά μας. Και ισχύει το εξής, η ψηφιακή βιομηχανική πολιτική στις κορεσμένες αγορές ε, οι παίκτες είναι γνωστοί εδώ και δεκαετίες. Bayer, ABB, Airbus, ε, βιομηχανία Peugeot, Fiat, BMW, Nestlé ή αν θέλετε η Siemens, GE, Philips, iStorm και πολλοί άλλοι. iStorm και πολλοί άλλοι. Στον ε, ψηφιακό τομέα αυτές οι εταιρείε ε, γεννήθηκαν μόλις πριν από 20 χρόνια Γι' αυτή λοιπόν μια startup στην Κοπεχάγη, στο Παρίσι, στο Μιλάνο, στο Λονδίνο, στη Ρήγα, στο Βίλνιου, στο Ταλίν, στη Μαντρίτη. Γιατί αυτές οι νεοφύης επιχειρήσεις μετά από 10 χρόνια να μην έχουν επικρατήσει στην αγορά με τις δικές τους ιδέες και τις πλατφόρμες. Η Nokia, ας πούμε, πριν από 5 χρόνια είχε το 50% της αγοράς στα κινητά τηλέφωνα και σήμερα μηδέν. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει και η αντίστροφη εξέλιξη. Εγώ είμαι πεπισμένος για αυτήν και πάνω σε αυτήν πρέπει να δουλέψουμε. Η κυβερνοασφάλεια, ναι, αλλά και τα G4, τα G5, είμαι υπέρ της ε, επικοινωνίας με G4 και G5 και είμαι και ε, σαφώς υπέρ ε, της χρηματοδότησης μέσα του προγράμματος Horizon 2020. στις, ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε στον ψηφιακό κόσμο ε, ως την άλλη πλευρά, όχι απαραίτητα ως εχθρό, να δεχόμαστε τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς στο θέμα της ουδετερότητας του διαδικτύου να δέχεται τις ΗΠΑ και από την άλλη να θέλει να καταστρέψουμε το Google δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτά που λέει ο Ομπάμα σχετικά με την ουδετερότητα των δικτύων ε, και ούτε να θέλουμε η Κομισιό να καταστρέψει το Google ή το ένα ή το άλλο. Εγώ είμαι υπέρ ε, του μέσου δρόμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εταίροι συν ε, ε, ε, και η Google είναι ευπρόσδεκτη στην Ευρώπη. Όμως η Google οφείλει να δέχεται τις δικές μας τις ρυθμίσεις περί κοινής αγοράς, το δίκαιό μας περί ανταγωνισμού. Και ε, Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν 80 ενστάσεις από επιχειρήσεις στην Ευρώπη και χαίρομαι που η παλιά επιτροπή δεν κατέληξε σε απόφαση και η πρόταση ε, για ε, οδηγία του περασμένου έτους απορρίφθηκε. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε να υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία θα διαφυλάσει την απαραίτητη ουδετερότητα και αντικειμενικότητα. Η μηχανή αναζήτησης να μην προτιμάει τα δικά τα προϊόντα και να είναι ε, με διακριτική μεταχείριση έναντι των άλλων. Ο ψηφιακός κόσμος δεν πρέπει να έχει διακρίσεις και αυτές είναι οι προσδοκίες μας έναντι της Google και εφόσον τις ικανοποιεί κανένα πρόβλημα. Αν ε, όχι, ελπίζω να αναζητήσουμε κάποια λύση. Και ένα άλλο παράδειγμα. Σήμερα το πρωί διάβασα ότι η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων λόγω νομικών γνωμοδοτήσεων του Πανεπιστημίου της Λουβέν ε, και των Βρυξελών λέει ότι ε, αυτή αυτές οι οδηγίες χρήσης ε, που εφαρμόζει το Facebook εδώ και ένα χρόνο δεν συμβαδίζουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ε, θα το ελέγξουμε και αν ισχύει αυτό για το Facebook θα βγάλουμε όχι μόνο την κίτρινη αλλά και την κόκκινη κάρτα στο Facebook. Εγώ δεν είμαι κατά του Facebook αλλά όπως λειτουργεί στον ευρωπαϊκό χώρο με δεδομένα θα πρέπει να σέβεται τους δικούς μας τους κανόνες. Αλλιώς ε, θα λάβει κυρώσεις ή θα τον πετάξουμε έξω. Αυτό αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Όχι ε, με χθρότητα απέναντι στις ΗΠΑ, στη Μουμπάη, στη Σανγκάη, στο Πεκίνο ή πουδήποτε αλλού, ούτε και απέναντι στο Τόκιο. Και το τελευταίο που θέλω να πω σχετικά με την ουδετερότητα του δικτύου. Ε, κοιτάξτε, δεν έχω δεσμευτεί. Γνωρίζω όμως και θέλω να πω το εξή. Αν τελικά καταλήξουμε σε κάποια οδηγία, χρειαζόμαστε την ε, έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και οι δύο θα πρέπει να κουνηθούν. Ε, και τους καλώ να δείξουν κάποια χαλαρή διάθεση να μην βάλουν τη ζώνη ασφαλείας και να παραμείνουν ακούνητοι. Στο Συμβούλιο λοιπόν η ουδετερότητα του διαδικτύου δεν ταυτίζεται με αυτό που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας το επισημαίνω. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω. Όταν με ρώτησαν κατά πόσον δίνω προτεραιότητα ε, σε ε, υπηρεσίες διάσωσης ε, ή στους αναλυτές τραπεζών, που δεν είδε δίνω προτεραιότητα στους αναλυτές τραπεζών. Αν οι υπηρεσίες διάσωσης μπορούν να δείξουν, να αποδείξουν ότι μπορούν να σώσουν ζωές, τους προτιμώ προφανώς σε οποιαδήποτε περίπτωση. Και αν πιστεύουμε στην κινητικότητα και αν το αυτοκίνητο ε, τα επόμενα 10 χρόνια θα παίζει κάποιο ρόλο ε, στις ευρωπαϊκές μεταφορές και μπορούμε να αποδείξουμε ότι η αυτοματοποιημένη οδήγηση μπορεί να οδηγήσει στον να αποφευθεί τον 90% όλων των θανάσιμων και μη ε, ατυχημάτων τότε προφανώς θα έχει προτεραιότητα στο διαδίκτυο. Άρα δηλαδή απαντάτε εδώ και το ερώτημα ότι αν μπορούν να περιστούν τα τροχαία θανατηφόρα ατυχήματα, προφανώς και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από τους αναλυτές των ε, τραπεζών ή τους πολιτικούς. Λυπάμαι, μακάβριο είχε αυτό, αλλά εγώ έτσι ε, αντιμετωπίζω τη ζωή. Αυτό σημαίνει ρεαλισμός. Και αν έχουμε ε, στην επαρχία ένα νοσοκομείο με 80 κλίνες που δεν είναι όμως αποτελεσματικό, αλλά με αυτό προσφέρεται κάποια υπηρεσία. Αυτό δεν μπορεί να κλείσει και εκεί ακόμα κι αν ένας από τροχαίο τύχημα ε, κινδυνεύει να πεθάνει και μπορεί να ε, θεραπευτεί, να χειρουργηθεί μάλλον σε μισή ώρα γιατί αλλιώ θα πεθάνει και δεν υπάρχει εκεί κανένας ε, γιατρός γιατί αυτός πάει στην πανεπιστημιακή κλινική που είναι μακριά 100 χιλιόμετρα αν μπορεί όμως αυτός ο γιατρός να χειρουργήσει ψηφιακά, δηλαδή πώς σε πραγματικό χρόνο να δίνει εικόνες στον επιτόπου γιατρό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και άρα διατηρείται το επαρχιακό νοσοκομείο, αλλά αυτός όμως, σας λέω, έχει ψηφιακή κάλυψη για περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από το να έχουμε μουσική που να την κατεβάζουμε από το YouTube ή να παίζουμε παιχνίδια ή να ε, μεταφέρεται το ποδοσφαιρικό αγώνα Νίρεμβέργης κατά Στουτγάρντης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ήταν πολύ μακροσκελής η να παιζουμε παιχνιδια η να μεταφερεται το ποδοσφαιρικο αγωνα νιρεμβεργης κατα Στουτγάρτη. ευχαριστω πολυ κυριε επιτροπε ηταν πολυ μακροσκελης η απαντηση σας, πλήρης. Έχω άλλους 15 συναδέλφους στο κατάλογο δεν μπορείτε να μιλήσετε ούτω ή άλλω πάνω από 1,5 λεπτό καθένα. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τρία λεπτά θα μιλήσω ο επίτροπο στο τέλος. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουν και οι 15 συνάδελφοι και να πούν την άποψή του επί του ζητήματος. Η κυρία Αλτερελ Καστίγιο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί είμαστε πολλοί και το θέμα είναι σαφώς σημαντικό και ιδιαίτερα δελεαστικό. Ε, δεν είναι μόνο σημαντικό. Πρώτον, πρέπει να υπενθυμίσουμε τον τίτλο, το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου σε σχέση με τους προηγούμενους Επιτρόπους. Είναι Επίτροπος για την, οικονομία και την, ε, ψηφιακή οικονομία και ψηφιακή κοινωνία. Επομένως, δεσμεύεται από τις αρμοδιότητές του με την Επιτροπή μας κυρίως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε λίγο να καθορίσουμε ότι ο πυρήνας των αρμοδιοτήτων σε αυτή την ενιαία ψηφιακή αγορά είναι αδιαμφισβήτητα της Επιτροπής Ήτρε. Και αυτό φυσικά ε, είναι γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων και των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν τρία πράγματα. Πρώτον, για το είναι ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, για την DSM, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και εδώ συμφωνώ με τον Επίτροπο, διότι κατά την άποψή μου υπάρχει τουλάχιστον μια ευκαιρία με τη Λετωνική Προεδρία να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ουσιαστική συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί στη διάρκεια αυτή τη προεδρία, αλλά ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ε, μετά από τις προσπάθειες της Ιταλικής Προεδρίας που έκανε καλέ προσπάθειες, αλλά δεν κατάφερε να έχει μια ε, κοινή θέση το Συμβούλιο. Θεωρώ όμω ότι βρισκόμαστε πλέον ε, πολύ κοντά στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Σαφώ αυτή η κοινή θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το φάσμα, το ουδετερότητα του δικτύου και την περιαγωγή διαφέρει από αυτή του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου, αλλά εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μια διαδικασία συναπόφασης, που σημαίνει ότι όπως και εμεί ε, τροποποιούμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση κανονισμού, ε, αντίστοιχα θα πρέπει τελικά να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι αποτέλεσμα των αρχικών μας θέσεων ε, και μία απόπειρα στη συνέχεια να βρούμε μία συμφωνία η οποία θα είναι επαρκώς ικανοποιητική. Δεύτερε, Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη πολύ σύντομα γιατί ήθελα να πω και κάτι ακόμα διότι δεν έχω άλλο τρόπο. Ε, ένα ακόμα πράγμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Επίτροπε, ότι ακόμα το ψηφιακό θεματολόγιο έχει ξεκινήσει. Είχε ξεκινήσει για το 2020 και ε, είμαστε στο 2015. Ε, άρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όσον αφορά την παρακολούθηση ε, για να δούμε αν ισχύουν κάποια πράγματα, αν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πλέον δεν ισχύουν, δεν ισχύουν, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία τη εφαρμογή του ψηφιακού θυμολογίου. Θα μπορούσατε να μα πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα του άξονε που θα περιλαμβάνει η ανακοίνωση για την ψηφιακή αγορά, την οποία περιμένουμε ε, προσεχώ από το Συμβούλιο, είπε ο Ευχαριστώ. Καταλαβαίνετε ότι είστε αρμόδια, ε, καταλαβαίνω ότι είστε αρμόδια για τον τριμερή διάλογο, γι' αυτό σα άφησα να επεκταθείτε λίγο περαιτέρω, αλλά σα παρακαλώ συνάδελφοι να τηρείτε το χρόνο. 1,5 λεπτό. Ο κύριο Σταγιάννη, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Γκούντερ, για την απάντησή σου για την Google. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Χρειαζόμαστε ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην Ευρώπη για την περιαγωγή. Τι άποψη έχεις για μια διπλή στρατηγική, μια διτή προσέγγιση, να εντοπίσουμε τα προσκόμματα και να τα άρουμε αργότερα. Για τις υποδομές. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερα για τις ψηφιακές υποδομές, χρειαζόμαστε περισσότερα ευρωπαϊκά ψηφιακά προγράμματα και θα πρέπει να ενώσουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά όχι μόνο με το σχέδιο επενδύσεων Juncker, αλλά και με την ε, ε, ε, Ένωση των Κεφαλαγορών για να έχουμε κατάλληλη χρηματοδότηση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις μας. Και θα ήθελα, Γκούντερ, να σε ρωτήσω. Σκοπεύεις να δημιουργήσεις στενό σύνδεσμο μεταξύ της ε, ε, νέας ψηφιακής αγοράς και της FinTech για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά και εντός χρόνου. Μπράβο, μπράβο. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Συμφωνώ κύριε Επίτροπε, με αυτά που είπατε σχετικά με την επιτάχυνση της νομοθετικής μας εργασίας. Απαραίτητο αυτό και χαίρομαι που λέτε ότι αυτό το κάνει τώρα το Συμβουλίο στο πακέτο των τηλεπικοινωνιών. Ε, εμείς ε, στο Κοινοβούλιο, ήδη κατά την προηγούμενη θητεία, είχαμε καταθέσει προτάσεις με τη βοήθεια των εισηγητών και σκιωδών εισηγητών. Τώρα όμως το ρόλο να λαμβάνει το Συμβούλιο και αυτό πρέπει να επιδείξει ευελιξία έτσι ώστε επιτέλους να εγκριθεί αυτή η δέσμη μέτρων. Σας στηρίζω λοιπόν. Δεύτερον, Όσον αφορά το δίκαιο περί δικαιωμάτων δημιουργού, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό που έχει σημασία στο νέο copyright να υπάρχει μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στους διάφορους εμπλεκόμενους. Πολίτες, ε, δημιουργούς και τους αποκαλούμενους ενδιάμεσους. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε αυτή την οικονομική αλυσίδα. Εχθές ε, είχαμε μια μακρά συζήτηση ε, για την έκθεση RAID Πρόκειται για την εφαρμογή εφαρμογή της παλιάς οδηγίας copyright. Εκεί συζητήσαμε σε βάθος και θέλω να σας ενημερώσω ότι σχεδόν όλοι όσοι ζήτησαν το λόγο υπογράμμισαν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τους δημιουργούς μας ε, στην Ευρώπη. Ε, τους ε, λογοτέχνες, συγγραφείς, όλους εκείνους. Αυτό είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας και αν δεν κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, τους προστατεύσουμε με το copyright. Ε, αυτό δεν μπορεί να θέλουμε να ε, τους αφήσουμε εκτεθειμένους. Όλοι συμφωνούμε από αυτό και σας τα λέω αυτά γιατί ε, έγινε συζήτηση η συνάδελφη που κατέθεσε την πρόταση δίνει σημασία μόνο στους χρήστες και δεν συμφωνήσαμε επ' αυτού εχθές στην Επιτροπή. Ο κύριος Ζωρίνιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την υποστήριξή μου για την ψηφιακή ένωση. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Απαραίτητο να καταλήξουμε σε μια κοινή στρατηγική για τον τομέα αυτό. Ορισμένοι θεωρούν και βλέπουν το ψηφιακό θεματολόγιο απλώς ως εργαλείο, ως μέσο βελτίωσης μιας υφιστάμενης κατάστασης. Όμως κατά την άποψή μου το ψηφιακό θεματολόγιο δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτό. Είναι ένας τρόπος, ένα μέσο για να ε, βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Να, παρέχει, να παρέχουν εταιρείε που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες και πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Κατακτώντας μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς. ένα είδος ευρωπαϊκού Silicon Valley, αν θέλετε. Μπορεί να ξεκίνησε το ίντερνετ από την Αμερική, αλλά δεν χρειάζεται να παραμείνει η Αμερική στην πρώτη θέση. Πρέπει λοιπόν να άρουμε τα εμπόδια που υπάρχουν. Χρειάζεται μεγαλύτερη, μεγαλύτερη, περισσότερες επενδύσεις, χρειάζεται περισσότερη καινοτομία, περισσότερη έρευνα Και αυτό είναι ο μόνος τρόπος να μην μείνουμε πίσω σε σχέση με άλλε περιοχέ του κόσμου, με άλλε χώρε του κόσμου. Αύριο, κύριε Επίτροπο, όπω γνωρίζετε, αναμένουμε την ε, ανακοίνωση για την Ενεργειακή Ένωση. Και το ερώτημα είναι πότε εσεί θα κάνετε τη δική σα ανακοίνωση για την Ψηφιακή Ένωση. Ευχαριστούμε, κυρία Κρίφιν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η βιομηχανία του θεάματος είναι ένα ε, στοιχείο κλειδί της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και μπορεί να αξιοποιήσει την ε, ψηφιακή ένωση για να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, το μοντέλο της πνευματικής ιδιοκτησίας που ακολουθούμε στην Ευρώπη φαίνεται να έχει μείνει στο 19ο αιώνα. Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο το οποίο να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιθυμίας των χρηστών περιεχομένου ταυτόχρονα προστατεύοντας τα συμφέροντα των υπολείπων που βρίσκονται στην αλυσίδα παραγωγής περιεχομένου, τους ε, δημιουργούς, τους ε, καλλιτέχνες, τους ε, εμπορευόμενους αυτό το περιεχόμενο επίσης. Σήμερα τα πνευματικά δικαιώματα περιορίζονται στο ποσό που πληρώνεται στον δημιουργό. Υπάρχουν όμως πλατφόρμες ε, ανταλλαγής τραγουδιών που, είναι, ε, που δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τα δικαιώματα του δημιουργού και μπορώ να σα δώσω παραδείγματα και από τη δική μου χώρα. Το ερώτημα είναι τι θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το κενό που υπάρχει και να διασφαλίσετε ότι τελικά οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες θα έχουν την ε, κατάλληλη σωστή αμοιβή για τη δουλειά τους. Υπάρχουν ε, εταιρείε των οποίων η έδρα μπορεί να βρίσκεται στις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά αξιοποιούν την ε, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, κρύβονται πίσω από αυτήν και στην πραγματικότητα υπονομεύουν τις ε, θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να υπάρχουν στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία, βρίσκεστε και από μια πόλη που μας δημιουργεί μια ζήλια αυτό. Έχω δύο ερωτήματα για τον... Ε, Σχετικά με το πρόγραμμα Juncker μιλήσατε ε, για το θέμα αυτό και ρωτώ. Τι είναι εκείνο που σας καθιστά αισιόδοξου ότι θα μπορούμε και από το πρόγραμμα Juncker να χρηματοδοτήσουμε τον ψηφιακό κόσμο. Αν αφαιρέσουμε δηλαδή την Connecting Facility ή ε, σε σχέση με κάποιες άλλες δυνατότητες του Horizon 2020. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Εσείς συμφωνείτε στο πλαίσιο του προγράμματος Juncker να έχουμε ως προτεραιότητα και την ε, πολιτιστική και ε, δημιουργική κοινότητα της Ευρώπης. Γιατί αυτό είδαμε δυστυχώς ότι δεν είναι προτεραιότητα. Το τρίτο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Είπατε ότι πρέπει να επιταχύνουμε ε, παρουσιάσατε τη βραδίτα που υπάρχει. Η οδηγία NIS είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Είναι μια παραδοσιακή συζήτηση όπως γίνεται και στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Βεβαίως οι Αμερικανοί που όλοι τους βρίζουν, οι Αμερικανοί μέσα από τον έλεγχο του χρηματιστηρίου εξέδωσαν μία απόφαση όπου με βάση την οποία οι επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο χρηματιστήριο μπορούν να αναφέρουν στους ισολογισμούς τους ζημιά που υπέστησαν από hackers. Αυτό τώρα λοιπόν δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Ξέρετε όμως κάτι, οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, να αποκαλύπτουν απώλεια δεδομένων και πολλά παρεμφερή. Γιατί αυτό δεν το θεωρείτε ότι είναι παράδειγμα, ότι δεν πρέπει να προχωράμε παραδοσιακά, αλλά θα πρέπει με μεγαλύτερη ενέργεια να αντιμετωπίζουμε θέματα ρύθμισης και αποφάσεων που μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τον παραδοσιακό νομοθετικό τομέα. Ο κύριος Κάλεϊ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Με χαρά σας άκουσα στις σημερινές σας παρουσίες όπως και κατά το παρελθόν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συμφωνήσω με όλα όσα είπε ο συνάδελφος και με κάλυψε κιόλα. σε σχέση με το φάσμα. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτών που προτείνεται στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Και αναφερθήκατε επίσης στο roaming, στην περιαγωγή. Υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του 2015 θα καταργούνταν πλήρως οι χρεώσεις για το roaming. Θα ισχύει αυτό ή εγκαταλείψαμε αυτή την ιδέα επίσης. Όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και τις επιθέσεις, το hacking, ε, είμαστε 10 χρόνια πίσω. Και το ερώτημα είναι μπορούμε να κινηθούμε όσο γρήγορα χρειάζεται για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Και σε αυτή την περίπτωση ε, τα μέτρα που θα λάβουμε για την κυβερνοασφάλεια τι επιπτώσεις θα έχουν στην, ε, στο ανοιχτό ίντερνετ και την ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ που θα θέλαμε να έχουμε. τη ελευθερία που θα θέλαμε να έχουν οι πολίτες να μπορούν να σερφάρουν στο ίντερνετ και να χρησιμοποιούν δεδομένα. Τώρα, εάν... Θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει με το δίκτυο για τα υφή οχήματα, γιατί αν κάποιος καταφέρει να παραβιάσει αυτό το σύστημα θα δημιουργήσει χάος στο δικό δίκτυο. Ευχαριστούμε κυρία Σάντερς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Έτιγκερ για το γεγονό ότι εξέφρασε την, ε, το ενδιαφέρον του για τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα και βρίσκουμε, έρχομαι από την ε, Αλσατία έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι περνούν τα, σύνορα κάθε μέρα για να εργαστούν στην Γερμανία. Επομένως ε, τα, τα, τα τέλη για το roaming είναι κάτι το οποίο μου διαμαρτύρονται συστηματικά. Τα τέλη πυραγωγής λοιπόν, κύριε Επίτροπε, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι συγκεκριμένα η πρόταση, η, η πρόβλεψή σας, τι πρόκειται να γίνει με το θέμα αυτό συγκεκριμένα. Δεύτερο ζήτημα. Επενδύσεις για την ανάπτυξη της ψηφιακή κοινωνίας. Προφανώς χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο. Κατάλληλο. Χρειάζονται επίση υποδομέ, χρειάζονται επίση κεφάλαια, το είπαν και οι συνάδελφοι. Αλλά επίση νομίζω χρειάζεται και μια διαφορετική νοοτροπία. Μιλάμε συχνά για την επιχειρηματική νοοτροπία που χρειάζεται για να ξεκινήσει κάποιο μια εταιρεία, αλλά εγώ επίση αναρωτιέμαι πώ μπορούμε να ενισχύσουμε ε, μια ψηφιακή, αν θέλετε, φιλοσοφία, νοοτροπία στου επιχειρηματίε που ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και γενικότερα στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, παρουσιάσετε νομίζω με διαφάνεια το κατάλογο των εμποδίων που αντιμετωπίζουμε στη δημιουργία της ψηφιακής ένωσης. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτόν τον κατάλογο. Είναι η πολύ μεγάλη διαφορά που υπάρχει, το χάσμα που υπάρχει τι ψηφιακέ δεξιότητε ανάμεσα στι διαφορετικέ ομάδε του πληθυσμού. Γι' αυτό οδηγεί τελικά σε διακρίσει, οδηγεί σε αποκλεισμό ε, των πιο ηλικιωμένων ή ατόμων στι αγροτικέ περιοχέ. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε την ψηφιακή οικονομία, την ψηφιακή κοινωνία, αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και αν δεν φροντίσουμε οι ψηφιακέ δεξιότητε κάθε πολίτη να βελτιώνονται. Ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Κάτι ακόμα. Ε, κύριε Επιτροπή, υπάρχει ένα μυστικό που θα ήθελα να μας αποκαλύψετε. Έχει σχέση με την TTIP. Τι προβλέπετε στην TTIP, ή στις για την TTIP, όσον αφορά την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και την, ε, ελεύθερη, την ελευθερία πρόσβασης ε, των ατόμων στην ψηφιακή ανάπτυξη. Κυρία Τόγια, κύριε Επίτροπε, εκτιμώ ιδιαίτερα το αίτημά σα να υπάρχει δεύτερη εντολή διαπραγμάτευση για το ραδιοφάσμα. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει ε, να παρετηθούμε ενώπιον τη αδυναμία ή τη μη βούληση του Συμβουλίου να επιλύσει το ζήτημα και όπω λέγατε και εσεί εδώ και καιρό στο Κοινοβούλιο συζητάτε αυτή η πτυχή και υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να λάβουμε υπόψη. Υπάρχει προστιθέμενη αξία αν υπάρχει πιο συντονισμένη άποψη για το ραδιοφάσμα διαμεθοριακά. Ε, και το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο πολλοί μειοδοτικοί διαγωνισμοί ε, ε, αφορά όχι μόνο την οικονομική κατάσταση αλλά και το πώς αντιμετωπίζεται το θέμα στις διάφορες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό και από τεχνικής και από οικονομικής αλλά και πολιτικής πλευράς να εμβαθύνουμε στο θέμα του ραδιοφάσματος και χαίρομαι που ζητάτε μια δεύτερη διαπραγματευτική εντολή. Όσον αφορά την αιρετερότητα του δικτύου, εγώ δεν κατάλαβα το παράδειγμα που μας κάνατε. Μας κάνατε παραδείγματα για την οδική ασφάλεια, για τις πρώτες βοήθειες, για την αυτόματη οδήγηση. Αυτά όλα εντάσσονται σε όλη αυτή τη ε, συζήτηση της καθολικής υπηρεσία ή τη Υπηρεσία κοινή ωφελία. Εμείς δεν θέλουμε ισότιμους όρους επ' αυτού για την ουδετερότητα του δικτύου. Εμείς αναφερόμαστε στις υπηρεσίες που πολλούνται. Πολλούνται ω ειδικέ υπηρεσίες όταν στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν ε, νέα τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα στο διαδίκτυο τα παραδείγματα τα οποία μας κάνετε σαφώς θα πρέπει να την χάνουν προτιμιασιακής ε, ε, μεταχείρισης και να αποτελούν προτεραιότητα, διότι πρόκειται για υπηρεσίες κοινή ωφελία. Ποιο μπορεί να αρνηθεί την προτεραιότητα στις πρώτες βοήθειες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ουδετερότητα του δικτύου δεν τίθεται και για τις υπηρεσίες, οι οποίες ε, πολλούνται με κάποιο αντίτιμο αρκετά υψηλείο. Και δεν κατάλαβα γιατί μας κάνατε αυτά τα παραδείγματα για την ουδετερότητα του δικτύου. Για την ε, περιαγωγή θα ήθελα να σας καλέσω να επιμείνετε, γιατί νομίζω ότι θα είναι και διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τριμερή διάλογο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια και δίνουμε μάχη από αυτού. Ευχαριστώ, ο κύριος Φανίστερ Λόι, στη συνέχεια. Πολύ σύντομα. Τέθηκαν ερωτήσεις ε, για τις υποδομές και τις πραγματικές επενδύσεις και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχετε κάποια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε ιδιωτικό κεφάλαιο για επενδύσεις. Υπάρχει ε, η δυνατότητα Connecting Europe που πήγε από τα 20 δις στο 1 δις και υπάρχει και το επενδυτικό σχέδιο Juncker τώρα. Έχετε κάποια ανάλυση, κάποια εικόνα για το ποιες είναι οι δυνατότητές μας εδώ. Τα πάντα θα χρηματοδοτηθούν μέσω πιστώσεων, οι οποίες πρέπει να αποπληρωθούν. Ε, θεωρώ ότι με το νέο δίκτυο θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ένα ε, μοντέλο και να το επανεξετάσουμε. Έχετε κάποια στοιχεία, έχετε πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επ' αυτού. Ευχαριστώ κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Ετυγκό, η βιομηχανία έχει, η ευφυής βιομηχανία έχει γίνει της μόδας η ολοκληρωμένη βιομηχανία και ε, αυτή η διασύνδεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία μοιάζει να είναι ως μοναδική ευκαιρία για την οικοδομική ανησυγκρότηση της Ευρώπης. Το ότι εσείς αποδίδετε σημασία στο θέμα αυτό φαίνεται και από το ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ε, διάσκεψης που οργανώνεται για τους stakeholders το αφιερώνεται σε αυτό το θέμα. Αν όμως το δούμε πιο προσεκτικά θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις για να υπάρξει τομή σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, καταρχήν, να υπάρχει μια εκτεταμένη ευρυζωνικότητα, εμπιστοσύνη στα δεδομένα και ενιαία γλώσσα. Δηλαδή, σαφής ορισμός των ενιών, έτσι ώστε σε τελική ανάλυση, ανεξάρτητα ποιο θα είναι ο κατασκευαστής, οι μηχανές, οι συσκευές να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα δύο πρώτα που έθιξα υπάρχουν στο πρόγραμμα Juncker ή αν θέλετε στα προγράμματα για την μεταρρύθμιση της προστασίας των δομένων και της προστασίας των εργαζομένων. Όχι όμως το τρίτο. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει η Ευρώπη έτσι ώστε να ενισχύσει αυτό το θέμα στο πλαίσιο της βιομηχανίας 4 προς 0. Of course, we are short of time, you see it. Δεν έχουμε χρόνο. Έπρεπε να είχαμε τελειώσει πριν από πέντε λεπτά. Αλλά και ο Επίτροπος δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις διεξοδικά, αλλά θα μπορούσαμε να σας ζητήσουμε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα, να, σας, να έρθετε στην επόμενη συνεδρίαση. Είναι απολύτως απαραίτητο να συζητηθεί περαιτέρω το ζήτημα. Αν θα μπορούσατε λοιπόν να μας κάνετε αυτή την παραχώρηση, και να κάνετε τώρα μια τελική δήλωση, κύριε Επίτροπη, γιατί πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και σίγουρα θα σας ξανακαλέσουμε στο εγγύς μέλλον, σε μελλοντική συνεδρίαση. Λοιπόν, για το πρόγραμμα Juncker. Δώστε μας λιγάκι κάποιες εβδομάδες, κάντε υπομονή έτσι ώστε οι γενικές διευθύνσεις και ο συνάδελφος κ. Κατάινεν να καταλήξουν στα καλύτερα κριτήρια για τη μόχλευση της ψηφιακής υποδομή. Και βέβαια πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι κάνουν οι προπολογισμοί των κρατών μελών, των περιφερειών, ε, των δήμων και κοινοτήτων και τι κάνει η τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία. Πρόκειται για δισεκατομμύρια, υπάρχει ανάγκη επενδύσεων πολλών δισεκατομμυρίων και κυρίως ε, στις ε, επαρχίες χωρίς μόχλευση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Διότι ο αριθμός των πελατών ε, και ο κύκλος εργασιών για τα επόμενα χρόνια δεν φτάνουν. Όσον αφορά τώρα την ε, ψηφιακή εσωτερική αγορά. Ο να Αντσιπούν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι ε, θα καταθέσουν το σχετικό πακέτο το Μάιο. Ε, θα συμμετέχει και η Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης, αυτή για ανταγωνισμού, για θέματα βιομηχανίας, ο Επίτροπος για θέματα πολιτισμού, ο υποφαινόμενος και ε, όλοι και εγώ υποφαινόμενος ε, το Μάιο ε, θα σας παρουσιάσουμε τις συζητήσεις για τις διάφορες ψηφίδες του, της δέσμης μέτρων. Η οδηγία NIS είναι πολύ σημαντική για μας για την ευρωπαϊκή προστασία δεδομένων. Ελέγχθησαν διάφορα και εγώ τα προσυπογράφω συμφωνώ και επαυξάνω. Ε, πρόκειται μόνο για μία πλατφόρμα, για μία πρώτη δέσμη μέτρων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, ε, και μετά πρέπει να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό πολιτισμό, ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ασφάλεια των δεδομένων. Στην ευρωπαϊκή βιομηχανία έχουμε πολύ καλές επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν τις τεχνικές δυνατότητες για να υπάρχει μεγαλύτερη ε, ασφάλεια δεδομένων. Και θεωρώ ότι εδώ υπάρχει και μια πολύ καλή ευκαιρία για, ε, για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αναφερθήκατε στην Αλσατία. Κοιτάξτε, πράγματι η ε, δομή των υποδομή δεδομένων δεν παραμένει και δεν σταματάει στα σύνορα. Ε, ας πούμε, ο Χασάπης, με ο Κρεοπόλης στο Στρασβούργο που έχει τη δυνατότητα να προμηθεύει κάποιον στο μέλλον αδρυμό, ε, θα παίρνει με ψηφιακό τρόπο παραγγελίες, συμπληρωματικές παραγγελίες και όλα αυτά θα πρέπει να είναι σε πραγματικό χρόνο, όχι με καθυστέρηση ημερών. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε διασυνοριακά την ίδια ταχύτητα, την ίδια ποιότητα των δικτύων μας, παράλληλη εξέλιξη σε οικονομικούς χώρους, οι οποίοι σαφώς και είναι σε διαφορετικές χώρες. Ας πούμε για την πυριαγωγή, όταν τηλεφωνείτε από το Στρασβούργο προς τον Μπορντό, αυτό είναι πολύ πιο φθηνό από ότι από το Στρασβούργο στο Κέλ. Μα το Κέλ είναι πολύ πιο κοντά στο Στρασβούργο. Ε, και το λειτουργικό κόστος είναι πολύ πιο μικρό από ότι να τηλεφωνεί κανεί από το Στρασβούργο στο Μπορντό. Γι' αυτό λοιπόν οι επιχειρήσεις ε, τηλεπικοινωνικές καταλαβαίνουν την όλη προβληματική της ε, περιαγωγής. Άρα δηλαδή πρέπει το στομότερο δυνατόν να ρυθμιστούν τα θέματα με την οδηγία TSN και εγώ βασίζομαι στο ότι η απόφαση του Κοινοβουλίου ε, θα είναι ικανοποιητική με βάση την πρόταση του Συμβουλίου. Το τελευταίο, η βιομηχανία και τα δίκτυα καθιστούν απαραίτητο να χρησιμοποιούμε και να ορίσουμε τις λέξεις και τη γλώσσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο έτσι θα μπορεί κανείς να συνονοηθεί. Υπάρχουν βέβαια οι αρμόδιοι φορείς ε, της ε, τυποποίησης. Αυτοί πρέπει να το πράξουν, διότι χρειαζόμαστε σε πραγματικό χρόνο όχι μόνο την ίδια υποδομή, αλλά και την ίδια γλώσσα, εφόσον μιλάμε για επικοινωνία μηχανών ανάμεσά τους και για ε, αυτόματη επικοινωνία βιομηχανικών μονάδων. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπετε ότι δεν μπόρεσε ο Πίτροπος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας αναλυτικά, αλλά προσπάθησε τα έχει σημειώσει τα υπόλοιπα ε, και θα τις θυμάται και θα τις επαναλάβει ε, τις απαντήσεις την επόμενη φορά ε, στο εγγύς μέλλον. Θα τον καλήσουμε γιατί θέλει να έχει καλές επαφές, συνεχείς επαφές και να έχουμε μια καλή αντιλογή απόψεων. Η συζήτηση αυτή ήταν διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξεκινάμε κάτι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Πίτροπε. Ναι, ε, ε, Συνάδελφοι, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ένα πολύ σημαντικό σημείο, αναφέρθηκε και από τον Επίτροπο Έτιγκερ πριν από λίγα λεπτά, το σχέδιο επενδύσεων Juncker, ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου. Θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο κάτι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για μια πρόκειτη ανταλλαγή απόψεων. Βιαζόμαστε σε αυτή την περίπτωση, διότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τα πάντα και τον τριμερή διάλογο τον Ιούνιο. Επομένως, σε τέσσερις μήνες. Αλλά στην επόμενη σύνοδο στο Στρασβούργο θα ε, γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Ήτρε ε, στη Δευτέρα στις 9 Μαρτίου 7.30 με 9.30 δύο ώρες αφιερωμένες αποκλειστικά στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δύο ώρες συζήτηση. Δευτέρα βράδυ, Στρασβούργο. Και την επόμενη μέρα επιπλέον, την Τρίτη δηλαδή στις 10 Μαρτίου, 5.30 με 7.30 το απόγευμα, 5.30 με 7.30 άλλες δύο ώρες για το θέμα αυτό άτυπη συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρε με τον Αντιπρόεδρο Κατάινε και τον Επίτροπο Μουέντας. Και οι δύο θα είναι παρόντες. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, Παρασκευή 13 Μαρτίου. Μπορεί να μην αρκεί ο χρόνος με αλλά θα τα καταφέρουμε. Σήμερα θα θέλαμε ε, η συνεδρίασή μας να διαρθρωθεί ως εξή. Να ακούσουμε τον εισηγητή, την άποψή του και τους κοιόδης εισηγητές, ίσως και τους συντονιστές σε κάποιες περιπτώσεις, για κάποιες μικρές παρεμβάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για σήμερα, να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και να ακούσουμε τι έχουν να πούν ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές. Και επίσης να ξέρουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό και όπως βλέπετε έχουμε 35, ίσως και 40 λεπτά στη διάθεσή μας. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Κατλίν Βαμπρέντ, η οποία είναι η συγχύτρια. Έχετε πέντε λεπτά. Πόσα? Πέντε. Πέντε. Εντάξει κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ πολύ που ανακοινώσατε και τι άλλε δυνατότητε έχουμε να συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να παρέμβουν όλοι. Οι προθεσμίε πραγματικά μα πιέζουν, ακόμα και εμένα ως εισηγήτρια, δεν έχω ακόμα την έκθεση. Ακόμα ε, είμαι στη διαδικασία... Ε, ανταλλαγής απόψεων και αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, είναι πολύ σημαντική. Θα υπάρξουν αρκετέ διμερές συναντήσει τι επόμενε ημέρε, ώστε να έχουμε μια καλή βάση. Καταρχάς ε, θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς, ελπίζω να μπορώ να μιλώ ε, εξ ονόματος της Επιτροπής, καλωσορίζουμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ε, ζητήσαμε μια πληρέστερη και βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική επενδύσεων εδώ και αρκετό καιρό. Και ε, έπρεπε να αλλάξουμε από την ε, ε, λιτότητα στις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Και αυτό φυσικά αποτελεί μια πρώτη αρχή. Ίσως είναι λίγα και κατόπιν εορτής, αλλά να σας πω ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ τουλάχιστον να προσπαθήσουμε εμείς από πλευράς της Επιτροπής μας αυτό το επενδυτικό σχέδιο να μην χάσει από την εκκίνηση. Και αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτά τα λίγα λεπτά είναι να σας παρουσιάσω μια εικόνα αυτών που θεωρώ εγώ ότι είναι τα τρία βασικά στοιχεία για την Επιτροπή μας. Εμείς είμαστε η Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί ε, για το άρθρο 54, επομένως υπάρχει ε, αποκλειστική αρμοδιότητα και τουλάχιστον στην αρχική μου έκθεση θα επικεντρωθώ σε αυτή την αποκλειστική αρμοδιότητα. Υπάρχουν άλλες ε, επιτροπές που έχουν άλλες αρμοδιότητες για να ασχοληθούν με αυτό το δύσκολο θέμα, σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ε, κατά την άποψή μου, τα ουσιαστικά στοιχεία είναι τα εξή. Καταρχά, ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση του σχεδίου Juncker θα γίνει με τα χρήματα που ε, λαμβάνονται από το ΟΕΣΔΑ 2020, που ήταν πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας, αλλά και από το Connecting Europe, που είναι ένα σημαντικό τμήμα της ε, χρηματοδότησης των ενεργειακών υποδομών, και αυτά τα κονδύλια δεν θα επηρεάσουν ή θα επηρεάσουν όσο το δυνατόν λιγότερο την ε, ακαιρεότητα του θεματολογίου για την ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία. Δεύτερον, να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα και οι εγγυήσει του Ταμείου θα χρησιμοποιηθούν σωστά. Δηλαδή η επένδυση απλώς και μόνο δεν αρκεί. Θα πρέπει να δούμε τι, πού και πότε θα επενδύσουμε. Οι επιπλέον επενδύσεις, οι επενδύσεις οι οποίες αλλιώς δεν θα υλοποιούνται, επενδύσεις οι οποίες όχι μόνο δημιουργούν οικονομικό αντιστάθμισμα, αλλά και ένα αντιστάθμισμα για την κοινωνία. Θέσεις εργασίας, επενδύσεις στην πραγματική περιφερειακή οικονομία και φυσικά ε, την περιβαλλοντική και ενεργειακή ατζέντα μας. Και τρίτον, να διασφαλίσουμε ότι η διακυβέρνηση των ταμείων θα εγγυάται πλήρη εφαρμογή των μέσων και συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο. Δηλαδή, δεν πετάμε τα χρήματά μας απλώς σε ένα ταμείο χωρίς να έχουμε κανέναν έλεγχο στη συνέχεια για το τι θα γίνει. Να περάσω τώρα στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που έχω όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι πολύ σημαντικό να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να τεθούν πριν ε, περάσουμε στην εκπόνηση της έκθεσης και στην κατάθεση των τροπολογιών. Από πού προέρχονται τα κονδύλια. Το Κοινοβούλιο, και νομίζω ότι δεν ήμουν μόνο εγώ, και άλλοι ευρωβουλευτές ε, ήταν εδώ στην Επιτροπή που εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά για να υπάρχει μια ισορροπία στον ορίζοντα 2020. Μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ του κλάδου, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ερευνητικών κινητήτων, ε, τα κράτη-μέλη, τις εθνικές πλατφόρμες. Μια πάρα πολύ δύσκολη ισορροπία και με ανησυχεί πάρα πολύ σήμερα και νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι και εδώ στην αίθουσα ανησυχούν, ε, διότι η ισορροπία που καταφέραμε να επιτύχουμε τώρα διαλύεται με, την, ε, με τον νέο κανονισμό. Είναι λογικό, για παράδειγμα, να υπάρχει μια νέα ανακοίνωση για την Ενεργειακή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα οι απαραίτητε επενδύσει που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτή τη Ένωση, ε, για παράδειγμα, για καλύτερη διασύνδεση, ε, εγκαταστάσει αποθήκευση κλπ., ε, δεν θα υλοποιηθούν, θα παρακολουθούν. Θα ήθελα πραγματικά να δω τι γίνεται με την ισορροπία στο ορίζοντα 2020 και στο Connecting Europe. Επίσης, θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε και τη δυνατότητα εναλλακτικής χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα από το αποθεματικό ή άλλες τεχνικές προϋπολογισμού που είναι διαθέσιμες. Εγώ δεν είμαι ε, η δήμον σε θέματα προϋπολογισμών, ε, επομένως στρέφουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους που γνωρίζουν καλύτερα τα του προϋπολογισμού εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερα χρήματα από τον ορίζοντα 2020, ήδη θεωρώ ότι αυτό θα αποτελεί μεγάλη βελτίωση για Αυτού που εργάζονται στον τομέα αυτό που ανησυχούν ιδιαίτερα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τον ορίζοντα 2020 ή τμήμα του ορίζοντα 2020 και του Connecting Europe. Δεύτερον, τι συνέπειες θα υπάρχουν στις ε, ε, προτινόμενες περικοπές, στην αρχική ισορροπία και για τον ορίζοντα 2020 και το ε, Connecting Europe. Θα πάει στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, θα δημιουργήσει μόχλευση. Τρίτον, σχετικό με αυτό, πώς ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πώς να περοκόψει τον προπολογισμό του ορίζοντα 2020. Αν, για παράδειγμα, σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το επιχείρημα της μόχλευσης, πώς αιτιολογείται το γεγονός ότι ε, περικόπτονται, περικόπτονται δαπάνες από τη θεμελιώδη έρευνα που ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα τα ξαναδεί αυτά τα λεφτά, και δεν θα μπορέσουν φυσικά να ε, επωφεληθούν από το ημόχλευση στο στρατηγικό ταμείο. Και επίσης γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει το κεφάλαιο για την ε, ε ηγετική θέση της βιομηχανίας όταν ε, ασχολούνται πάρα πολύ στενά με τις αγοράς, ε, από, πολύ πιο στενά από τη θεμελιώδη έρευνα. Θα ήθελα να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα κατανομή για να έχουμε πάλι ισορροπία στους διάφορους τομείς στο ορίζοντα 2020. Δεύτερον, θα προσπαθήσω να τα πω λίγο πιο γρήγορα κύριε Πρόεδρε, από πού προέρχονται τα χρήματα και πώς μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό και πού θα πάνε. Η πρόταση για το Ταμείο Στρατηγικών Υποδέσεων λέει ότι η υποστήριξη της επενδύσης θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη και συνεχής ε, των στόχων της ε, πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μα, Αν δείτε τα διάφορα θέματα που μα ενδιαφέρουν, ε, ήταν εδώ μόλι ο επίτροπο για την Ψηφιακή Ένωση. Αν δείτε ε, τις ψηφιακέ υποδομές, τις μικρομεσαίες επιχειρήσει, εμεί είμαστε η Επιτροπή που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Καταρχά, τα επιπρόσθετα στοιχεία. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η υποστήριξη του στρατηγικού ταμείου δεν θα επενδύσει σε πράγματα τα οποία θα, στα οποία θα είχαμε επενδύσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, από τη μια θα έχουμε κοινωνικοποίηση του κινδύνου και ιδιωτικοποίηση ε, ε, της ε, επιβεβαίωση των τρεχόντων προγραμμάτων. Δεν θέλουμε να δώσουμε τα χρήματά μας εκεί λοιπόν. Και επίσης η συνέπεια με την ενωσιακή πολιτική. Κάτι το οποίο αναφέρεται σαφέστατα στο άρθρο 5, για το οποίο υπάρχει και πάλι αποκλειστική αρμοδιότητα στον προτινόμενο κανονισμό και θα ήθελα να αναφερθώ στην αλλαγή του κλίματος, στην περιβαλλοντική πολιτική, ε, νομικά δεσμευτικούς στόχους, ε, τους οποίους θα θέλαμε να έχουμε σε πιο φιλόδοξο επίπεδο, ε, η οδηγία για την ποιότητα του αέρα, το 7ο πρόγραμμα, το το 7ο συγγνώμη, πρόγραμμα δράση και ούτω καθεξή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει σαφής καθοδήγηση, κάπω να μπορέσουμε να περιχαρακώσουμε τα πράγματα, να υπάρχει κατάλληλη ανάθεση κολυνδυλίων, ώστε να ξέρουμε ότι τα χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα ε, είναι επένδυση σε όλου αυτού του τομεί. Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο, στη διακυβέρνηση, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για την Επιτροπή μα και για άλλε επιτροπέ. Η ε, Διευθύνουσα Επιτροπή και Επιτροπή Επενδύσεων του Στρατηγικού Ταμείου, ιδίω η δεύτερη, θα πρέπει να έχει κατάλληλο τρόπο ελέγχου των μέσων που διευθύνεται και θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι εμπειρογνώμονε που θα συμμετέχουν. Είναι ε, από διάφορου τομεί, ε, μπορούν να κάνουν αξιολογήσει οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ για του σαφεί μα στόχου. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να συμμετέχει ιδιαίτερα στον έλεγχο της εφαρμογής του Στρατηγικού Ταμείου και μια φορά το χρόνο να έρχονται εδώ στην, Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή μας για ε, να δίνουν λόγο δεν αρκεί. Ε, υπάρχουν ε, προηγούμενες εμπειρίες από προγράμματα για την έρευνα, καινοτομία, για ε, τις υποδομές της των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών και πρέπει να φροντίσουμε η διακυβέρνηση του Στρατηγικού Ταμείου από τη μια να λειτουργεί και αυτό φυσικά δεν επαφείται σε εμά, ε, δεν θα αποφασίζουμε εμείς για το κάθε πρόγραμμα, αλλά πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε ότι οι προτεραιότητές μας είναι αυτές που πρέπει να είναι και λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστώ. You see it was not so bad. Ευχαριστώ, είδατε. θα καταφέρατε σε μόλις 9 λεπτά. Δεν τηρήσατε ακριβώ το χρόνο, αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον η παρέμβασή σας. Πάντω ήταν απολύτως απαραίτητο να πείτε όλα αυτά που είπατε. Είμαι βέβαιο ότι θα μπορούσατε να την πει ακόμα περισσότερα. Ε, ε, ζητώ συγγνώμη τώρα για τα ε, περιορισμούς που σας θέτω, αλλά υπάρχουν τυπικοί περιορισμοί και η Επιτροπή ε, προπολογισμού και η ε, Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιε, με βάση τον κανονισμό άρθρο 55. Εμεί περιοριζόμαστε στο άρθρο 18, 19, δηλαδή στα άρθρα για τον ορίζοντα 2020 και, τους, και, το Connecting Europe, το συνδέοντα στην Ευρώπη. Θέλω να συμφωνήσω με τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμουμε τη ε, εξέταση του άρθρου 19, γιατί και οι δύο επιτροπές, και η δική μας και η ΤΡΑΝ, είναι αρμόδιες για το άρθρο 19 και για τους στόχους του EFSI, αυτού του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Ταμείου Επενδύσεων, είναι το ερώτημα που έθιξε και η συγγήτρια, τι θέλουμε τελικά. Για τα επόμενα δύο χρόνια οι στόχοι που θα τεθούν θα είναι πολύ σημαντικοί. Αυτό από την πλευρά των, τύπων. Ξεκινώ για τους, με τους σκιώδες εκ μέρους του ΕΛΚ ο κύριος Έλερ, Πόσο να πούμε τώρα, είναι 2 και 10, 3 λεπτά ο καθένας παρακαλώ, 3 λεπτά οι σκιώδες. Μπορείτε. Κύριε και κύριοι, εκτός μικροφώνου. Having been the... Ήμουν σε συνεργασία με την Τερέζα Μοντρέλο, ε, συνεισηγητής η λογική της μόχλευσης που συχνά ακούγεται είναι το επιχείρημα ότι ας βρούμε μια επιδότηση, ας τη στείλουμε στη χρηματοοικονομική αγορά και αυτό θα οδηγήσει σε μόχλευση. Αυτό δεν ισχύει. Ένα εκατομμύριο που περικόπτουμε από τον ορίζοντα 2020 οδηγεί σε απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων από τον επιχειρηματικό τομέα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει κάτω το παρελθόν. Το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Juncker λοιπόν δεν θα επιτυχεί τους στόχους του εάν ακολουθήσουμε τη λογική που λέει ότι πρέπει να είναι σοσκελισμένα αυτά τα προγράμματα Αν ακολουθήσουμε λοιπόν τη λογική που λέει ότι θα χρειαστεί επένδυση από ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο στα προγράμματα αυτά. Το ζήτημα λοιπόν είναι επίση το εξή. Εάν έχουμε, το πολιτικό, εάν έχουμε μια περικοπή 7,2 δισεκατομμυρίων από τον ορίζοντα, αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα είχαν στη διάθεσή του τα χρήματα αυτά δεν θα το έχουν. Το ίδιο και τα ερευνητικά κέντρα, τα κέντρα αριστεία. Σε προγράμματα στα οποία συμμετείχαν πάνω από 7.000 μέλη του, επιχειρηματικού τομέα της βιομηχανίας. Ούτε αυτοί. Επίσης οι φοιτητέ. Επίσης οι ερευνητέ. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν επιπτώσεις αυτές οι περικοπές που κάνουμε στον ορίζοντα 2020. Και επί της ουσίας αυτό θα οδηγήσει σε περικοπές στις, στην καινοτομία στην Ευρώπη. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι μήπως υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις να αναζητήσουμε από αλλού χρηματοδότηση και κατά την άποψή μας ναι υπάρχουν. Υπάρχουν αποθεματικά, υπάρχουν τα διαφορετικά ταμεία, υπάρχει διαθέσιμο χρήμα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ήταν η εύκολη λύση να πούμε ότι την ερευνητικό προϋπολογισμό μπορούμε να κόψουμε, δεν τους νοιάζει και πολύ. Όταν το 80% των βραβευθέντων με βραβείο Νόμπελ που βρίσκονται εν ζωή απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του ζητούν να μην προχωρήσει σε αυτέ τι περικοπέ για την έρευνα, πρέπει να του λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Εάν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, πρέπει να βεβαιωθούμε, πρέπει να, να μας εξηγήσει κάποιος ποια θα είναι η διαφορά. Επίσης, ζητούμε μια διάμεση αξιολόγηση όλα τα χρηματοδοτικά μέσα που έχει εγκρίνει ποτέ το Κοινοβούλιο προέβλεπαν μια διάμεση αξιολόγηση. Γιατί είναι εύκολο να ε, γίνει μια αρχική κατανομή, αλλά να διαπιστώσουμε μετά από στη μέση του δρόμου ότι 400 εκατομμύρια ευρώ τελικά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, για παράδειγμα. Και επίσης, είχαν εδώ επίτροπος και μας είπε ότι στον τομέα της ψηφιακής υποδομής, δώστε μας λίγο περισσότερο χρόνο, 4-6 εβδομάδες, για να καταλάβουμε ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα. Και αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ της, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, του Ευρωπαϊκού, και, και, συγγνώμη, και της βιομηχανίας, από τις οποίες έχει αποκοπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς λοιπόν αυτές οι συζητήσεις μπορούν να αντακατοπριστούν στην νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νομοθετική πρόταση. Η ουσία της όποιας πρότασης πρέπει να βρίσκεται στην νομοθετική πρόταση. Η δεύτερη επιλογή, δεύτερη όμως επιμένω επιλογή είναι η πράξεις κατεξοδότηση και λέω ότι είναι δεύτερη επιλογή γιατί αυτές αποκόπτουν λίγες από τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου τις ελεκτικές. Συμφωνούμε ότι πρέπει να ορίσουμε τις προτεραιότητες και ότι η αρμοδιότητα για τον ορισμό των προτεραιοτήτων βαρύνει τις επιτροπές μας με βάση το άρθρο 55. Επίσης. Δεν θέλουμε να αποκόψουμε χρήματα από άλλα ταμεία ή από τον ορίζοντα, το ορίζοντα 2020. Και βλέπετε ότι το σημαντικό στοιχείο είναι η λεπτομέρεια σε αυτών των προγραμμάτων. Το είδαμε και χτες. Και έχει πολύ ενδιαφέρον που συζητούμε μεταξύ μας για τα μέλη της Επιτροπής Οίκων και Προϋπολογισμού, Οικονομικών Θεμάτων και Προϋπολογισμού. Αναφερόμαστε σε αυτή την ξανθιά κυρία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από αυτήν την πρόταση, εάν δεν την δούμε ολοκληρωμένη και δεν δούμε τις λεπτομέρειές της, εκεί μόνο θα καταλάβουμε αν μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από τα χρηματοδοτικά μέσα που ήδη υπάρχουν. Για αυτό το ζήτημα που θέσατε με τους συναδέλφους θα το συζητήσουμε μετά. Ο κύριος Γκρομπάτσικ. Και εγώ θα εστιάσω στις λεπτομέρειες που λέτε. Χρειάζεται επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης, λέμε όλοι, συμφωνούμε σε αυτό, ιδιαίτερα για να ξαναυπάρξει μια ισορροπία, για να δημιουργηθεί μάλλον μια ισορροπία ανάμεσα στην ε, Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη και να σταματήσει η μετανάστευση από την Ανατολή προς τη Δύση. Γι' αυτό χρειάζεται να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα τη βαριά βιομηχανία, την πληροφορική, την, ε, μεταφορές την αυτιλία και οπουδήποτε μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεύτερον, χρειάζεται να αποκτήσουμε ενεργειακή ανεξαρτησία, αυτονομία. Αυτό είναι απαραίτητο για την Ευρώπη για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική όταν υπάρχει μια φτηνή πηγή ενέργειας σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να την αξιοποιεί τόπου. κάτι που θα διασφαλίσει και την ανεξαρτησία μας από τους παρόχους ενέργειας που βρίσκονται στην Ανατολή και γενικότερα από άλλους, άλλες χώρες στον κόσμο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντεμπάκερ, εκ μέρους της Άλντε. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, όπως και δύο προλαλήσαντες, θα ήθελα να μάλλον θα ήθελα να συμφωνήσω με του δύο προλαλήσαντε σε σχέση με την ανάλυση που κάνουν. Πρώτα απ' όλα, από πού θα έρθουν τα χρήματα. Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι έχει υπάρξει μια πολιτική απόφαση η Επιτροπή να επιλέξει να βρει τα χρήματα από εκείνα τα ταμεία που θεωρούσαν ότι δεν θα δημιουργήσουν πολιτικέ αντιδράσει. Είναι η εύκολη λύση, αλλά είναι η βελτιστή. Κατά πάση πιθανότητα όχι. Είπε και ο συνάδελφο από το ΕΛΚΟ ότι υπάρχουν και αλλού αποθεματικά, ίσω από αλλού θα μπορούσαμε να βρούμε κονδύλια, αντί να κόψουμε το 20% του προπολογισμού που απευθυνόταν στην έρευνα και ήταν το μόνο μέρο του ευρωπαϊκού προπολογισμού που θα πήγαινε στην έρευνα. Μήπω λοιπόν καλύτερα να βρούμε άλλε πηγέ και να κρατήσουμε το, ε, το ε, SEF και τον ορίζοντα 2006, 2020, ε, με συγχωρείτε, ανέπαθο. Το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο θα είναι υπεύθυνο για την κατανομή αυτών των κοντιλίων, ποιο θα εφαρμόσει αυτήν τη στρατηγική. Η Τράπεζα Επενδύσεων φαίνεται ότι θα είναι εκείνη που θα είναι αρμόδια, αλλά με πιο ζήτημα διακυβέρνηση, το οποίο θα εξασφαλίσει ότι τελικά τα χρήματα αυτά θα φτάσουν στην πραγματική οικονομία. Θα συνεργαστεί με του φορεί επιτόπου τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τους, ε, τα πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά κέντρα επιτόπου. Ποιος θα έχει τη γνώση αυτή για να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία και να φτάσουν τα χρήματα αυτά εκεί που πρέπει. Καθώς επίσης και πώ θα φροντίσουμε οι ιδιώτε επενδυτέ οι οποίοι γνωρίζουν την κατάσταση επιτόπου να συμμετάσχουν. Δεν είναι δυνατόν οι αποφάσει αυτέ να ληφθούν στι Βρυξέλλε, στο Λονδίνο από μακριά εξ αποστάσεω. Χρειάζεται συμμετοχή του τοπικού παράγοντα. Με τον ορίζοντα 2020 με την... δημιουργήσαμε τη στρατηγική για την ε, έρευνα. Με το Connecting Europe, με το Συνδέοντα στην Ευρώπη, δημιουργήσαμε τη στρατηγική για τι τηλεπικοινωνίε και τα δίκτυα. Γιατί να ξεκινήσουμε από την αρχή. Επομένω, αυτά τα δύο χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να τα προστατεύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί εάν αρχίσουμε να απορροφούμε κονδύλια από αυτά και να τα ε, μεταφέρουμε αλλού, θα πρέπει να βρούμε πώ θα γίνει η μόχλευση. Και εγώ δεν έχω πιστεί ακόμα πώ μπορεί να γίνει αυτό. Πώ μπορεί να πάρουμε χρήματα τα οποία αρχικά προορίζονταν για ε, επιδοτήσει βασική έρευνα να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς για δημιουργία θέσεων εργασία. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Πώ λοιπόν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσει ότι θα υπάρχει επαρκή λογοδοσία, επαρκή έλεγχο αυτή τη στρατηγική και τη υλοποίηση τη. Χρειάζεται ε, και η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και η Ήτρε να ασχοληθούν με το θέμα ακόμα πιο επισταμένα. Άλλο ερώτημα. Είναι δυνατόν ε, οι κληρωμές να γίνονται σταδιακά, βηματικά, με δόσεις και όχι με καταποκοπήν ποσά έτσι ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και να μπορεί να λειτουργήσει και στην πράξη η ενδιάμεση αξιολόγηση. Τέλος. Ποια θα είναι η στρατηγική του ιδίου του Ταμείου. Πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, δημιουργήσουμε υπερβολικά σφιχτό πλαίσιο, αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κατευθυντηρίε αρχέ. Χρειάζεται να ε, χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία έχουν μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τα οποία μπορούν να παρακολουθηθεί η πορεία του και στα οποία να υπάρχει ιδιωτική επένδυση και να μην υπάρχει ψηλό βαθμό ρίσκου. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και ε, κάποιο ρίσκο, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα να χρηματοδοτεί κανεί μόνο σίγουρα προγράμματα. Επομένω, συμφωνώ με του συναδέλφου που λένε ότι τι λεπτομέρειε πρέπει να προσέξουμε. Εκεί θα, κάνουμε, θα, θα γίνει, βρίσκεται η διαφορά. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώ μπορεί αυτό το πρόγραμμα να εφαρμοστεί στο πεδίο και χωρί να ε, υπονομεύσει ή να δημιουργήσει προβλήματα σε επενδυτικά σχέδια που είχαν ήδη ξεκινήσει. Και να μην υπονομεύσουμε την ιδιωτική επένδυση, κάτι που συμβαίνει ήδη σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να διακόψω τη συζήτηση. Έχει σπάσει βέβαια το χρονόμετρό μας για να δω και πόσο μιλάτε. Ε, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε και μεγαλύτερες επενδύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό να το λέμε. Ε, λοιπόν, θα κοιτάω μόνος μου το χρόνο, θα σας σταματάω μετά από τρία περίπου λεπτά. Συνάδελφος Τούρμες, επόμενος μιλητής. Μ' αρέσει πάρα πολύ που δεν έχει κανείς από τον εφιάλτη του ρολογιού όταν μιλάει. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι βέβαια από πού προέρχονται τα χρήματα και εμείς είμαστε εκείνοι που θα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει ε, στις ε, διαπραγματεύσεις για την έρευνα. Δυόμιση χρόνια θέλαμε για να διαπραγματευτούμε ε, και κατά κάποιο τρόπο σιωπηρά τα μισά καταστράφηκαν. Και όπως είπε και ο Κρίστιαν, αυτό που ενδιαφέρει είναι η, η πραγματική καινοτομία στην Ευρώπη. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια έτσι ώστε να είναι σαφές και για τους επενδυτές ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, να είναι σαφής η ευρωπαϊκή υπεραξία και επίση, ε, κατά κάποιον τρόπο πρέπει να ε, προστατεύουμε τα επενδυτικά εργαλεία όπως είναι το Enofin. γιατί δεν έχει νόημα να σκοτώσει, να εξαφανίσει κανείς αυτό το εργαλείο. Ήδη έχουμε έξι χρόνια εμπειρίας και πολλοί λένε ότι θα προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα. Κατλίν, πράγματι εγώ συμφωνώ, χρειαζόμαστε έτσι μια περιχαράκωση και αυτή να συνδέεται και με κάτι άλλο που είναι πολύ κοντά σε αυτά που λέμε. Σε τελική ανάλυση οι, προ... οι προτάσεις και τα προγράμματα που θα κατατεθούν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνική αρρωγή. Άρα δηλαδή ε, το θέμα είναι τα χρήματα για την τεχνική αρρωγή θα διοχετεύονται σε ένα φορέα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή μήπως θα υπάρχουν και χρήματα για, τις τα πανεπιστήμια, ένα είδος ε, επιχειρηματικού κεφαλαίου για να βοηθηθούν και αυτά η τεχνική αρρωγή θα είναι αντικείμενο διαχείρισης μόνο κεντρικά. Για μένα λοιπόν υπάρχουν δύο πράγματα για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε την περιχαράκωση και χρειαζόμαστε επίσης να διασφαλίσουμε ότι ένα κομμάτι των κοντιλίων για την τεχνική αρρωγή θα δαπανώνται και εκτός ε, της κεντρικής αυτής δομής. Ναι, να υπάρχει κεντρική δομή αλλά και αποκέντρωση παραδείγματο για να βοηθηθούν οι πόλεις να μπορούν να ε, ξετυλίξουν τα μεγάλα τους προγράμματα και τα να μετατρέψουν σε προγράμματα επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τράπεζες. Ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα, ποια είναι η στρατηγική της Επιτροπής. Νομίζω ότι η πολιτική στρατηγική είναι εύκολο να γίνει κατανοητή. Δηλαδή θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Σήμερα κάποιος από την Επιτροπή μου είπε ότι το Συμβούλιο είναι κοντά στο να κλείσουμε συμφωνία. Και μετά η δεύτερη στρατηγική είναι ότι εδώ ε, θέλουν να κλείσουν συμφωνία με την Επιτροπή Προπολογισμών, όχι με εμά, γιατί γνωρίζουν ότι αυτή είναι κατά κάποιον τρόπο ανοιχτή πιο εύκολο να διαπραγματευτούν με εκείνους παρά με εμάς. Ε, το ε, τακτικής φύσεως πρόβλημα που έχουμε και αυτό μας αφορά όλους ε, είναι ότι οι δικές μας οι προθεσμίες ε, ε, για τροπολογίες είναι πολύ αργά. Δηλαδή η Επιτροπή ήδη κλείνει συμφωνία με τα κράτη-μέλη και μέσα από αυτή τη συμφωνία θα αυτήν μάλλον θα την επιβάλλουν στην Επιτροπή Προπολογισμών. Εμείς θα επεξεργαστούμε όλες τις λεπτομέρειες και μετά θα είναι πια πολύ αργά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει ε, να συντονιστούμε κάπως σε αυτό το θέμα και μέσα από τη γραμματεία πρέπει να σκεφτούμε το κατά πόσον μήπως η προθεσμία που προτείνουμε είναι πολύ αργά αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Συνάδελφος Φερέιρα, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω κατέστη σαφές από προηγούμενους ομιλητές, από τον εισηγητή και από τους σκιώδεις ότι εδώ έχουμε πάρα πολλές ε, επιφυλάξεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συνέχεια ίδιες επιφυλάξεις. Η συγγήτρια ε, στην αρχική της παρέμβαση τα εξήγησε όλα πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι το εξής. Από πού προέρχονται τα χρήματα και οι περιορισμοί ε, τα 2,7 δις έχουν επιπτώσει προφανώς. Εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε διοχετευτεί σωστά προς την κατεύθυνση της θεμελιώδους έρευνας. Ήταν περισσότερο στοχευμένο στις τελικές ε, φάσεις ε, της ε, έρευνας παρά στη θεμελιώδη έρευνα. Άρα δηλαδή η συμφωνία πλαίσιο, μάλλον οι περικοπές σημαίνουν ότι περισσότερα θα χάσει αυτή η θεμελιώδης έρευνα. Κάτι άλλο που μας απασχολεί είναι πού θα διοχετευτούν τα χρήματα και ποιος θα αποφασίζει για την κατανομή των κονδυλίων. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ. Και αυτό το ερώτημα θα το υποβάλουμε σε γραπτή μορφή ε, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Και κάτι άλλο, η σύνθεση του νέου ταμείου. Ε, θα έχουμε πολλές επιτροπές ε, ε, τελικά όμως ποιος θα αποφασίζει για τις ε, προτεραιότητες, ε, για την κατανομή των κονδυλίων και για το ποια προγράμματα θα χρηματοδοτούνται. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κανένας εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας, κανένας εμπειρογνώμονας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Άρα τελικά αυτοί οι εμπειρογνώμονες τίνο συμφέροντα θα υπερασπίζονται όταν θα φτάνουμε στο ερώτημα ποιος θα πάρει τα κονδύλια. Προφανώς και θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα εκείνων που θέλουν απόδοση, κέρδος από την επένδυσή τους ε, παρά τη μόχλευση. Όλα αυτά δεν είναι συμβατά με τα συμφέροντα που απορρέουν από άλλα προγράμματα που και αυτά τα δρομολογητούν. Άλλα προγράμματα θα παραμελητούν αν τελικά αυτοί οι εμπειρογνώμονες αποκτήσουν προτεραιότητα. Το θέμα είναι λοιπόν από πού θα έρθουν τα χρήματα, πώς θα δαπανηθούν και ποιος θα λαμβάνει τις αποφάσεις. Νομίζω είναι σαφές ότι η Επιτροπή Επενδύσεων και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι καθοριστική σημασία αυτού του θέματος. Ε, ξέρετε, το χρονόμετρο τελικά από ό,τι φαίνεται είχε σπάσει, ειδικά στη δική στην περίπτωση, τώρα δουλεύει μια χαρά. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε άλλον ένα συνάδελφο και τώρα κλείνει ο κατάλογος των ερωτώντων χωρίς να σας ρωτήσω. Και έχουμε ένα αίτημα προς τους διερμηνείς. Χρειαζόμαστε άλλα 10 λεπτά διερμηνίας και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μείνετε κοντά μας μέχρι τις 12.40. Ε, αλλά να είσαστε στην ώρα σας. Ομιλίες ενός λεπτού. Ο κύριος Συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν. Συμφωνώ, διότι υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Από πού προέρχονται αυτά τα κονδύλια και προς τα πού πάνε. Ε, ήμουν εισηγητής για το Connecting Europe Facility και τις τηλεπικοινωνίες ε, ε, από το ένα δις που είχαμε δώσει εκεί μένουν περίπου 200 εκατομμύρια και τα άλλα θα μεταφερθούν. Πού θα πάνε. Α, νομίζω ότι πρόκειται για ένα πολύ ε, εύλογο ερώτημα και είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά και συμφωνώ και με την εξή ανησυχία. Πώς ε, θα γίνει ο καθορισμός διότι για το Connecting Europe συζητούσαμε για πάνω από ένα χρόνο μέχρι να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία και τώρα πρέπει πολύ γρήγορα να καθορίσουμε τους κανόνες για το πώς θα βρεθούν φτάσουν τα χρήματα αυτά στο σύστημα. Πραγματικά λοιπόν τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά ε, γιατί είναι πολύ σημαντικές και οι επενδύσεις. Η κυρία Ουμπάτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιο ε, έθεσε μία ερώτηση για τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχει και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωράει στα τυφλά υπάρχουν ε, περικοπές στον προπολογισμό του ορίζοντα 2020, ενώ είναι ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως για τα ερευνητικά κέντρα. Είναι απαράδεκτο αυτό κατά την άποψή μου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την έρευνα, την καινοτομία, την παιδεία, τη δημιουργία μια σχέση μεταξύ των τριών και πάρα πολλέ χώρε έχουν πολύ συγκεκριμένα προγράμματα. Ε, και τα ερευνητικά κέντρα, για παράδειγμα, στον ορίζοντα 2020 θυσιάζονται. Και συμφωνώ με αυτό που είπε και η Κετλίν. Κατά την άποψή μου, το επίπεδο των περικοπών στη γραμμή προπολογισμών για τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Έρευνα και Καινοτομία θα πρέπει να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα είναι πολύ σοβαρές ανησυχίες που ελπίζω πραγματικά να τις διασκεδάσει κάποιος. Ε, πού πάνε και πού θα, από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια ότι δεν είναι δυνατόν να επενδύουμε σε ό,τι να είναι, γιατί σίγουρα με αυτό δεν θα πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Έχω και κάποιες επιπλέον ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με τα όσα ακούσαμε σήμερα. Και αυτό αφορά το πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν επενδύσεις βάσει των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και για το οι δέσμοι μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια του 2030 και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ε, θα χρηματοδοτούνται ε, ε, προγράμματα με ψηλό προφίλ κινδύνου σε σχέση με τα εφιστάμενα προγράμματα και πώς θα πάμε στη σωστή κατεύθυνση ώστε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να συνοδεύσουμε την αλλαγή για να έχουμε μια οικονομία χαμηλή σε άνθρακα. Ευχαριστώ κύριο Βανίστερλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τη θέση που ακολουθούμε είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η Επιτροπή προσπαθεί να αφουγκραστεί λίγο ε, ποιοι τομείς ε, θα είναι οι τομείς στους οποίους θα γίνουν περικοπές για να χρηματοδοτηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Και πολύ σωστά η εισηγήτρια έθεσε το ζήτημα. Γίνεται μια καλή συζήτηση. Καταφέραμε ε, μέσω της συζήτησης να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα του ορίζοντα 2020 και μπορεί ξαφνικά να έρχεται κάποιος και να κόβει ε, τα κονδύλια όταν έχει γίνει τόσο μεγάλη διαπραγμάτευση. Αν είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι είναι ισορροπημένο το όραμά μας, το, πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να δράσουμε ήδη εκ των προτέρων. Να μην περιμένουμε πάρα πολύ, να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τους συντονιστές για να προχωρήσει γρήγορα το θέμα. το προπολογισμό και το πού προέρχονται τα χρήματα είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους. Κύριε Τούρμε, θα διαβεβαιώ ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σκέφτεται πολύ σοβαρά από πού προέρχονται τα κονδύλια για τους αρχικούς στόχους που καθορίστηκαν στον προπολογισμό. Είναι αυτό το οποίο θέλει να περάσουν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς καμία τροπολογία και φυσικά δεν θέλουν να το συζητήσουν και μαζί μας. Εγώ δεν έχω ολοκληρώσει την εξέταση του ζητήματος, αλλά εάν προσπαθούμε να βρούμε από πού θα προέρθουν τα κονδύλια, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες εδώ για το ε, Connecting Europe. Για παράδειγμα, ο κύριος Έτιγκερ είπε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ιδιωτικά κονδύλια, ότι αυτά τα κονδύλια βρίσκονται στο Connecting Europe, για παράδειγμα για τις διασυνδέσεις του διαδικτύου και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να έχουμε κατάλληλες δομές για να υπάρχουν και υποδομές και να ε, δούμε λίγο και τι πολιτικούς στόχους είχαμε και πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτή θα είναι απόλυτα ε, σωστά στοχευμένοι. Στο 2020, στον ορίζοντα 2020, ε, κόβουμε τεράστια κονδύλια. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δουν και αυτά τι θα γίνουν. Ευχαριστώ, κυρία Έρνστα.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 ουσιαστικά τι κάνω, βγάζω από τη δεξιά τσέπη τα χρήματα που θα βάλω στην αριστερή τσέπη. Για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή η διαδικασία. Αν από τον ορίζοντα 2020, από το Connecting Europe ή από το αποθεματικό του προπολογισμού πάρω τα κονδύλια και τα βάλω σε άλλη γραμμή του προπολογισμού, ουσιαστικά είναι τα μόνα χρήματα τα οποία είναι εξασφαλισμένα. Όλα τα άλλα είναι λόγια, λόγια, λόγια και τίποτα άλλο. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αυτέ οι περικοπέ στον προπολογισμό ε, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα, τι ψυχία. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, ποιο ρόλο θέλουν να διαδραματίσουν όλα αυτά τα ζητήματα για το κλίμα, τις αποφάσεις που έχουμε γκρίνει εμείς, τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα ενεργειακά ζητήματα και ούτω καθεξής. Τι ρόλο έχουν να διαδραματίσουν όλα αυτά ε, τα προγράμματα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει άποψη σε αυτές τις τομείς ή είναι πράγματα τα οποία λέμε έτσι στον αέρα. Ποιος ε, ε, ελέγχει το Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων. Ποιο είναι λοιπόν αυτός ο οποίος τον ελέγχει. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο το κάνει αυτό και ε, πραγματικά έχω να εκφράσω πάρα πολλές αμφιβολίες από αυτό. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Σίγουρα είμαστε δυσαρεστημένοι γιατί πρέπει να αποφασίσουμε για τον ορίζοντα 2020 και το Connecting Europe. Ίσως ε, τόσο πολύ ε, για το Connecting Europe ε, όχι τόσο, αλλά τον ορίζοντα 2020 είναι πολύ σημαντικό. Και ως εισηγητή σε 7 θεμάτων κάποιες πρωτοβουλίες είναι πολύ καινούργιες. Για παράδειγμα το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, γιατί δεν είχε χρηματοδοτηθεί καθόλου στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χρηματοδότησης δεν θα χρηματοδοτούμε καινοτομία και τεχνολογία η αριστεία και η ευρύτερη συμμετοχή είναι επίσης μια νέα ιδέα. Η, η αδελφοποίηση και όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έπρεπε να απαντήσουμε σε όλα αυτά και τώρα πρέπει να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος James Hinton από την ΕΚΦΗΝ. Έχετε το λόγο, σας παρακαλώ δύο λεπτά και συγγνώμη γι' αυτό διαφορετικά ονομάζομαι Μελισσαράτο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είμαι σύντομο. Δύο ερωτήσει έχουν τεθεί. Από πού θα έρθουν τα χρήματα και πού πηγαίνουν. Από το πού προέρχονται. Καταλαβαίνω την κριτική η οποία ασκείται για τι περικοπέ που θα γίνουν στον ορίζοντα 2020 και το ΣΕΦ. Αλλά α μην ξεχνάμε τα ποσά για τα οποία μιλάμε. Πρόκειται για περικοπέ τι οποίε ορισμένοι χαρακτήρισαν δραματικέ κάθε άλλο εγώ θυμάμαι περίπου 79 δισεκατομμύρια τα επόμενα πέντε χρόνια και εδώ από αυτά τα 79 δισεκατομμύρια η περικοπή θα είναι 3,5. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δραματική περικοπή. Επίσης είπαν ορισμένοι ότι οι χρήματα τα οποία προεδι... πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επιδοτήσεις δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τις επενδύσεις. Αυτό πιστεύει και η Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι τα προγράμματα τα οποία προσφέρονται για επιδοτήσεις πρέπει να επιδοτούνται και τα προγράμματα τα οποία είναι επενδυτικά πρέπει να χρησιμοποιούμε κίνητρα για επενδύσεις. Για το ερώτημα λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και την επιθυμία του Κοινοβουλίου να υπάρξει λογοδοσία και έλεγχος αλλά χρειάζεται ε, και μια ε, ισορροπία. Γι' αυτό ζητούμε ανεξάρτητους εξωτερικούς ε, αξιολογητές. Χρειαζόμαστε προγράμματα τα οποία θα εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον και θα δημιουργούν θέσει εργασία, αλλά επίση πρέπει να είναι και στο χαρακτήρα του επενδυτικά. Άρα χρειαζόμαστε συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Αυτό είναι ουσιώδου σημασία στον τομέα αυτό. Και για να υπάρξει αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία, αυτή η συμμετοχή του ιδιωτικού παράγοντα, χρειάζεται ευελιξία. Άρα, καλή λογοδοσία, καλός ο έλεγχος, αλλά να μην φτάνουν οι όποιες αποφάσεις και κάθε φορά οι αποφάσεις να γίνονται πολιτικές, πολιτικού χαρακτήρα και να υπάρχουν πολιτικές αντεγκλήσεις. Γιατί αυτό θα αποθαρρύνει τους ιδιώτες επενδυτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, μην ξεχνάμε, την Τρίτη θα ζητήσω από την εισηγήτρια να κλείσει τη συζήτηση. Πάντως, πριν να σας ενημερώσω θα έχουμε δύο ώρε. συζήτηση με τον ε, Επίτροπο και τον Αντιπρόεδρο Κατάιναν για δύο ώρε στο Στρασβούργο. Και πριν θα έχουμε συζητήσει και μεταξύ μα. Η έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ όλου τους συναδέλφου και τους κοιόδες εισηγητέ και τους άλλου που πήραν το λόγο. Σε γενικές γραμμέ φαίνεται ότι συμφωνούμε. Έχουμε εντοπίσει όλα τα ίδια προβλήματα και η δουλειά μου τις επόμενες ημέρες είναι να κάνω διμερεί συναντήσει ή ομαδικέ συναντήσει ή οτιδήποτε άλλο για να ε, καταγράψουμε τελικά αυτή την κοινή θέση στην έκθεση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα σας αφουγκραστώ πολύ προσεκτικά και θα προσπαθήσω να συναντηθώ με όσου περισσότερου από εσά μπορώ. Ο πρόεδρο, ευχαριστούμε. Καλή τύχη, Κατρίν. Δεν είναι και εύκολο το έργο που αναλαμβάνει. Ε, Θα διακόψουμε τώρα τη συνεδρίασή μα και συνεχίζουμε στι 3. Ευχαριστά, ευχαριστεί ο Πρόεδρος και τους ε, διερμηνείς. Για αυτά τα 11 λεπτά παράτησης. Ευχαριστούμε. Καλό, καλή όρεξη.